Έχουμε μια πεφορτωμένη ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σα ζητήσω λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Προβλέπετε στην ημερήσια διάταξή μα καταρχήν μια ανταλλαγή απόψεων με τον Σέρβο Υπουργό Άμυνα, τον κύριο Ντράγκαν Σουτάνοβιτ, ο οποίο είναι δίπλα μου. Μετά με την κυρία Τζανέλα του Συμβουλίου για τα θέματα μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, τα θέματα του Ιράν, τα θέματα τη εξέταση από τη συνδιάσκεψη για τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων που έγινε τον προηγούμενο μήνα. Στη συνέχεια τη συζήτηση για το θέμα του Γαλιλαίου και την τροποποίηση του κανονισμού ο οποίος θεσπίζει ένα καθεστώς ελέγχου των εξαγωγών αγαθών διτής χρήσης. Είχαμε την ευκαιρία επίσης να έρθουμε σε επαφή με τους υπευθύνους της Αταλάντης, της Αταλάντας, του προγράμματος για την προστασία των ακτών της ε, Σομαλίας και επίσης είχαμε επαφή με την κοινοβουλευτή, είχαμε μια επίσκεψη στη Ρήγα στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ. Είμαστε στο διαδίκτυο, τρέχει, τρέχει η συνεδρία μας στο διαδίκτυο και μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ Άμυνα τη Σερβία. Καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία που έχουμε να σα συναντήσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε μαζί μα. Η Σερβία ακολουθεί το δρόμο της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο δρόμος της αυτός περνάει και από τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, ιδίως από τα θέματα ασφάλειας και άμυνας γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων οι χώρες αυτές ήταν στο παρελθόν καταναλωτές της ευρωπαϊκής ασφάλειας και τώρα γίνονται παραγωγή ασφάλειας, providers όπως λέμε στα αγγλικά και στην περίπτωση της Σερβίας είναι ακόμα πιο ευαίσθητο το θέμα αυτό γιατί όχι μόνο οι Σέρβοι ήταν μέσα εισαγωγικά καταναλωτές της ευρωπαϊκής ασφάλειας αλλά είχαν βρεθεί σε μια κάπως λεπτή θέση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εκ τούτου χαιρόμαστε που όλα αυτά είναι περασμένα ξεχασμένα και η Σερβία έχει μπει στον δρόμο αυτό του 21ου αιώνα και της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στη δική σας, στις δικές σας προσπάθειες, και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, η Σερβία έχει κάνει μερικές πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις ό,τι αφορά τις δυνάμεις ασφαλείας της και τις στρατιωτικές δυνάμεις της. Έχετε παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και πολιτικά για να βοηθήσετε όλη αυτή την περιοχή καθώς και τη χώρα σας για να εξασφαλίσετε μια μετριοπάθεια στις ενέργειες οι οποίες λαμβάνουν χώρο, να ζητήσετε να λάβουν χώρα διπλωματικές προσπάθειες και λύσεις και όχι στρατιωτικές ε, λύσεις που είχαν οδηγήσει σε γενικότερη ανάφλεξη στο παρελθόν. Εσείς παίξετε σημαντικό ρόλο και προσωπικά για τα θέματα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι έχει γυρίσει πλήρω η σελίδα σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, τις σχέσεις μα με τη Σερβία και όλοι μας θα πρέπει να θα από αυτό. Φυσικά παραμένουν κάποια θέματα τα οποία είναι ακόμα ένα ενεκρεμωτήτη. Η πρόθεση και η συμπλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Έχουμε πάντα ευαίσθητα θέματα όπως αυτά του κοσυφοπεδίου και μετόχια. Σας υπενθυμίζω ότι δεν είμαστε μαζί σας σήμερα για να συζητήσουμε το καθεστώς του κοσυφοπεδίου. Θέλουμε να μιλήσουμε για τον ευρωπαϊκό δρόμο της Σερβίας και ιδίως για αυτά τα οποία είναι στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και ιδίως για αυτά τα οποία εσείς προτίθεστε να κάνετε, δηλαδή το να ενταχθείτε στην κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σερβία είναι μία από τι τρίτε χώρε οι οποίε θέλουν να συνδεθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα αριθμό ενεργειών. Στα πλαίσια αυτή τη πολιτική, η διαπραγματεύση είναι εν εξελίξη και αυτό δείχνει ιδιαίτερα το πόσο ελκυστική είναι η πολιτική άμυνα και ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί τριτών χωρών. Αυτή η νέα εταιρική σχέση λοιπόν η οποία θα ξεκινήσει είναι ένα πολύ σημαντικό ε, στάδιο συνεργασία και πιστεύω θα αποδώσει και καρπού σε ό,τι αφορά την ένταξη της χώρας σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας αφήσω φυσικά το λόγο. Θα έχουμε και συζήτηση. Χαίρομαι επίση που είναι παρόν ο κύριος Κούκαν, ο οποίος προεδρεύει τι αντιπροσωπίε για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και έχουμε επίσης και τον κύριο Πάσκο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος αλλά αυτό είναι φυσιολογικό και ίσως είναι παρόν και ο κύριος <clears throat> Κατσίν, ο οποίο είναι ο εισηγητής για τη Σερβία και την κυρία Λούνα Τσέκ, η οποία είναι η αρμόδια εισηγήτρια για το Κωσικοπέδιο. Σας δίνω το λόγο κύριε Υπουργέ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να είμαι εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, πριν από δέκα χρόνια ήμουν ασκούμενος ε, και σαν κάποιους ε, που βρίσκονται σήμερα εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω. Το 2000 ήταν αυτό, όταν ο Μιλόσεβιτς στην εξουσία και δεν ήταν πολύ εύκολο να έρθω εδώ και να είμαι παρόν. Οπότε σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία για το μέλλον. Όταν μιλούμε για την ε, Σερβία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πω ότι για μένα πρώτη φορά, για, μένα το σημαντικότερο είναι καταρχάς ε, να, να γίνουν σεβαστές οι προδιαγραφές ε, στο Υπουργείο Άμυνας. Όταν μιλούμε λοιπόν για, τις, για τη μεταρρύθμιση, είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό αν δεν, γνωρίζουμε από πού ξεκίνησε κάνει, αν δεν γνωρίζουμε δηλαδή ποια, ήταν ε, η κληρονομιά μα ε, και πού βρισκόμαστε τώρα, από πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε. Είχαμε πλήρη έλλειψη κανονισμών ε, γιατί πριν από τις 15 Μαΐου Πριν από τις 15 Μαΐου είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με την έγκριση της μεταρρύθμισης αυτής. Είχαμε επίση πάρα, πολλά, πάρα πολλέ υποθέσει που εκκρεμούσαν ε, και στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Το 2005, από το 2005 έχουμε πάρα πολλέ υποθέσει που εκκρεμούν και έχουμε και μια πολύ κακή φήμη ως χώρα. Αρχίσαμε με την μεταρρύθμιση για την οποία σας ανέφερα επειδή είχαμε πάρα πολλά πράγματα στο πρόγραμμα μας πέρσι, εγκρίναμε και τους έξι νόμους ε, για το στρατό και την άμυνα. Έχουμε λοιπόν ένα νομοθετικό πλαίσιο και για πρώτη φορά επίσης εγκρίναμε μία εθνική στρατηγική για την άμυνα και μία έκθεση επίσης αναθεώρησης αυτής. Δεν ήταν βέβαια πάρα πολύ εύκολο αυτό. Ήταν, δεν ήταν εύκολο να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά επιτέλους καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτήν ε, την νομοθετική μεταρρύθμιση και από τον περασμένο Σεπτέμβρη έχει πλέον ολοκληρωθεί. Το 2007 τον Ιούνιο ολοκληρώσαμε και στο πλαίσιο του στρατού, στη διάρθρωση του στρατού ε, κάναμε μεταρρυθμίσεις ε, με προδιαγραφές ΝΑΤΟ, είναι ένας από τους καλύτερους στρατούς στον κόσμο και επίσης πρέπει να πω ότι έχουμε δημοκρατικό και πολιτικό έλεγχο στις στρατιωτικές μας, στις ένοπλες δυνάμεις, ε, και είναι κάτι το οποίο βέβαια έχει να κάνει και με την κατάσταση στο κοσυφοπέδιο ε, πολλές φορές είχαμε διπλωμάτες στη Σερβία που πολλές φορές μας ρωτούσαν ε, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε με αυτή την κατάσταση και αν ε, και, και η αντική μας απάντηση ήταν πάντα ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να κάνουμε κάτι που να αντίκειται στους νέους νόμους που προσπαθούμε να εγκρίνουμε. Βλέπετε και στη διαφάνεια ότι υπάρχει η πυραμίδα του στρατιωτικού επιτελείου Βλέπετε το 2005 είχαμε βλέπετε τον αριθμό των ε, διαφόρων ε, αντισυνταγματαρχών ε, και συνταγματαρχών. Βλέπετε επίσης ότι προσπαθήσαμε κάπως να αυξήσουμε το, την, το δημοφιλές ε, των ενόπλων ε, δυνάμεών μας, ε, να τις καταστήσουμε πιο αξιόπιστες και προσπαθήσαμε επίσης και τις στρατιωτικές ακαδημίες να εξυγχρονίσουμε. Φέτος είναι 129.000 ε, ε, που είναι ε, πολύ που είναι πολύ καλύτερα από το περσινό μας ποσοστό. Θέλουμε δηλαδή όλο και περισσότεροι νέοι να συμμετέχουν στις ένοπλες δυνάμεις. Επίσης βλέπετε ότι έχουμε πολύ καλά ποσοστά και, και στο πλαίσιο της ε, ε, κοινή γνώμης. Ε, έχουν γίνει σχετικές δημοσκοπήσεις. Είμαστε δεύτεροι στην εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης. Η πρώτη είναι η Εκκλησία. Την πρώτη θέση κατέχει η Εκκλησία στη Σερβία και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι γιατί προσπαθούμε να εξυγχρονιστούμε και αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ε, προς τις ένοπλες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, εκπονήσουμε οποιοδήποτε από τα καθήκοντά μας. Κάτι ακόμη που μας κάνει πολύ περήφανους Αναπτύξαμε πολύ καλές σχέσεις με πάνω από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, ειδικότερα στις, ε, με τις γείτονες χώρες πολλές συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας. Θα πάω και στο Ζάγκρεπ και θα υπογράψουμε συμφωνία και με το Ζάγκρεπ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι πολύ ευαίσθητη αυτή η συμφωνία και με όλες τις χώρες από την Άγκυρα μέχρι τη Βιέννη έχουμε σκοπό να υπογράψουμε τέτοιου είδους ε, συνεργασία ακόμη και με την Αλβανία. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα αυτών των συμφωνιών μας για να υπάρχει ε, συμφωνία των στρατιωτικών δυνάμεων της Σερβίας με όλες τις χώρες της περιοχής. Ε, Επίσης έχουμε, είμαστε πλήρες μέλος ε, στην περιφερειακή συνεργασία ε, των νοτιοδυτικών, ε, της νοτιοδυτικής Ευρώπης. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλες αυτές τις χώρες και επομένως δεν θεωρούμαστε χώρα που δημιουργεί προβλήματα όπως το παρελθόν. Ελπίζουμε να είμαστε πολύ πιο αξιόπιστοι και δεν, θα θέλα, δεν, δεν, δεν μπορούμε πια να κατηγορηθούμε ότι υποφάλπουμε κανέναν. Κάτι ακόμη που προσπαθούμε να επιλύσουμε για τα όπλα είχαμε περίπου 57.000 τόνους όπλων των οποίων ο κύκλος ζωής κλείνει, από υλικά των οποίων ο κύκλος ζωής κλείνει και μετά που μειώσαμε στους 17.000, ε, μειώνεται συνεχώς αυτός ο αριθμός και μάλιστα αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόβλημα και ζητούμε από τους φίλους μας και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθεί ε, το ε, νούμερο αυτό ακόμη περισσότερο. Δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, είναι πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής και προσπαθούμε να καταστρέψουμε τέτοιου είδους εξοπλισμό και προσπαθήσουμε να, προσπαθούμε μάλιστα να ε, εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας ε, γιατί είναι κάτι που αφορά όχι μόνο τη δική μας χώρα και άλλες χώρες. Ε, στο πλαίσιο τώρα των υποδομών ολοκληρώσαμε μία από τις μεγαλύτερες βάσεις στην Νότια Σερβία, πολύ ευαίσθητη περιοχή, σε πολύ ευαίσθητη περιοχή, λόγω των ε, μειονοτήτων που ζουν εκεί και προσπαθούμε να εξεύρουμε συμμάχους προκειμένου να υπάρχει μία ε, πολυτομεακή συνεργασία για την ενίσχυση της βάσης αυτής. Ε, περίπου 35 εκτάρια έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζουμε να φτάσουμε σε κάτι πάνω από 100 εκτάρια ώστε να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για τις ειρηνευτικές αποστελές, όχι μόνο για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις. Θέλουμε να ε, είμαστε πολύ πιο συνεργάσιμοι και με ε, ένοπλες δυνάμεις των γειτονικών χωρών. Όσον αφορά την KFOR τώρα, πρέπει να πω ότι η σχέση μας μαζί τους είναι πάρα πολύ καλή Είχαμε κάποια προβλήματα στο παρελθόν, αλλά πλέον δεν έχουμε προβλήματα, δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Ε, έχουμε σε τακτική βάση συνεργασία. Ο αρχηγός στρατηγού επιτελείου μας θα συναντηθεί με τον αρχηγό της ε, KFOR ε, αύριο και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό για μας. Επίσης υπάρχουν περιπολίες ε, για τις οποίες συνεργαζόμαστε, κάτι το οποίο σημαίνει πολύ μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ σερβικών δυνάμεων και KFOR. Είχαμε κάποια προβλήματα με τη μείωση του μεγέθους ε, στο Κωσυφοπέδιο και στα μετόχια, του μεγέθους των δυνάμεων της KFOR Δεν μπορώ να βρω την αγγλική λέξη, λέει ο μιλητής, μισό λεπτό. Προσπαθούμε να κάνουμε μια καλή ανάλυση για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των δυνάμεων ή όχι και σε τι βαθμό ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα στρατεύματα της ΚΕΙΦΟΡ. Είχαμε όμως κάποια προβλήματα μεταξύ των ε, ε, ε, Αλβανών και των Σέρβων Και από ό,τι άκουσα, ε, η Κέιφορ έκανε πολύ καλή δουλειά στο να προσπαθήσει να ηρεμήσει τα πνεύματα. Κάτι το οποίο κάναμε επίσης τα τελευταία τρία χρόνια. Είχαμε στρατεύματα σε ειρηνευτικέ αποστολέ ε, στη Λιβερία, στην ακτή ε, Ελεφαντοστού και στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στο Τσάντ Επίσης αποστήλαμε μια μεγάλη ατρική ομάδα στην περιοχή από πέρσι και την Πέμπτη εγκρίναμε μια κυβερνητική πρόταση για δύο ακόμη αποστολές στο Λίβανο και στην Κύπρο. Στο Λίβανο με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς και στην Κύπρο με τους Ούγγρους και τους Σλοβάκους φίλους μας. και ελπίζουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές στο μέλλον. Αυτό που επίσης μας ενδιαφέρει είναι να δούμε σε τι αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να συμμετέχουμε ώστε να είμαστε και εμείς παρόντες στις ε, ειρηνευτικές αυτές αποστολές. Τώρα, ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, για το επόμενο έτος. Το σημαντικότερό μας μέλημα είναι ο επαγγελματισμός ε, του ε, Σερβικού στρατού. Κατά την άποψή μου, αυτός είναι ο στόχος, ο μεγαλύτερος στόχος της ε, μεταρρύθμισης. Έχουμε ένα μεικτό σύστημα και μισθοφόρων και ιδιωτικής θητείας αλλά η υποχρεωτική στρατιωτική, θητεία θα καταργηθεί. 36.000 άτομα αριθμοί ο στρατός αυτή τη στιγμή. ...28.000 ε, στρατιώτες, ε, συν 2.000, ε, γιατί 2.000 άτομα θα είναι υπεύθυνοι εκπαίδευση των νέων στρατιωτών. Θα κάνουμε μια συμφωνία και με τους Κροάτες και τους Αλβανούς για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την περιφερειακή συνεργασία, πράγμα που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Ζούμε στον ίδιο χώρο από πλευράς ασφάλειας, από τα βόρεια ως τα ανατολικά, από τα νότια στα βόρεια, τα βόρεια στα δυτικά, τα δυτικά τα ανατολικά και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ασυμμετρικές απειλές όπως το διεθνές οργανωμένο έγκλημα δεν είναι απειλές μόναχα για μια χώρα, είναι απειλές για τη σύνολη περιοχή και πιστεύουμε ότι αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε καλές συνθήκες με τους εταίρους μας στις γειτονικέ χώρες μπορούμε να αποτρέψουμε τα προβλήματα αυτά. Έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή σε αποστολές διατήρησης της ειρήνης της, ε, του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια από τις πιο σημαντικές αποστολές για το Σερβικό στρατό. Έχουμε Έχουμε μια επιχείρηση διατήρηση της ειρήνης στο, στην Νότια Σερβία μαζί με μονάδες της K4. Θέλουμε παρόλα αυτά να συμμετάσχουμε και σε άλλους χώρους για να καταδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητές μας ασφαλείας και εκτός της Σερβίας. Το καλοκαίρι ελπίζουμε να ανοίξουμε ένα γραφείο εδώ στο αρχηγείο της, ε, του ΝΑΤΟ. Ο στρατηγός που είναι μαζί μου θα είναι ο εκπρόσωπός μας στο ΝΑΤΟ. Θα είμαστε λοιπόν οι καταναλωτές της διαδικασίας ασφάλειας όπως και οι άλλες χώρες θα έπρεπε ήδη να είχαμε ξεκινήσει από το 2006 που ήμασταν τμήματα της PFP, ε, της διαδικασίας. Αλλά είναι απαραίτητο να της ε, εταιρικής σχέσης για την ειρήνη, δηλαδή το PFP, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτές τις ιδέες. Έχουμε λοιπόν μια στενή σχέση με αυτές τις διαδικασίες αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε φυσικά προβλήματα και με τη χρηματοδότηση. Εμείς βάσει της κυβέρνησης της απόφασής μας θα έχουμε το 2,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για στρατιωτικούς ε, στόχους και για στρατιωτικές συντάξεις. Εφέτος πήραμε 2,12, είναι πολύ λιγότερο από ό,τι χρειαζόμαστε. Ελπίζουμε του χρόνου θα αυξηθεί η χρηματοδότηση αυτή για να προχωρήσουμε και στον εξυγχρονισμό του στρατού μας. Κάτι που είναι εξόχω σημαντικό για μας στο μέλλον. Μου είπατε 15 λεφτά, 15 λεφτά. μίλησα ως καλός στρατιωτικός και είμαι φυσικά έτοιμος να απαντήσω τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, δεν διευκρίνησα ότι όχι μόνο κάνατε ένα στάζ, μια μαθητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και ότι μετά την αλλαγή του καθεστώτος στο Βελιγράδι, Ήσασταν και στην ε, Επιτροπή Άμυνα του Κοινοβουλίου. Εδώ δηλαδή ακριβώ. Αυτή είναι εδώ την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Μα παρουσιάσατε μια πραγματικότητα πολύ σημαντική για όσοι παρακολουθούν τι εξελίξει ε, στα Βαλκάνια και στη Σερβία, όλο ιδιαίτερο. Μιλάτε για το μετασχηματισμό του στρατιωτικού μηχανισμού που ήταν ε, προβληματικός ε, μέσα στη δεκαετία του 90 και όπως υπενθυμίσατε είχε γίνει όχι μόνο για την περιοχή αλλά κυρίως για την ε, σερβική κοινωνία ε, έγινε τελικά ένα στοιχείο μια συνιστόσα ασταθερότητας για το σερβικό λαό. Τι άλλο πιο φιλόδοξο, πιο απαιτητικό να ζητήσουμε στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων της χώρας σας. Επίσης, συμμετέχετε στις ειρηνευτικές αποστολές της ΕΠΑ. Ξεκινάτε ένα κύκλο, ο οποίος θα συνεχίσει αύριο, ε, κύκλο προβληματισμού της Υποεπιτροπής ε, για τα, ε, Βαλκάνια. Ε, θα μιλήσουμε για την Αλτέα στη Βοσνία ε, και θα έρθουν διάφοροι εμπειρογνώμονες να μιλήσουν για τα θέματα των Βαλκανίων και κυρίως της Βοσνίας. Ο κύριος Πάσκου, ο αντιπρόεδρος Πάσκου. Ευχαριστώ. Σας χαιρετίζω. Είμαστε παλιοί φίλοι. Προσπαθούσα να κρυφτώ, αλλά με ανακαλύψατε. Βλέπετε που κάθομαι. Πριν ε, μπω μέσα, πριν κοιτάξω την οθόνη, έλεγα σε ένα φίλο ότι σας ήξερα πριν 10 χρόνια. 10 χρόνια νεότερος ήμουν τότε. Τότε αντιμετωπίσαμε κι εμείς παρόμοια προβλήματα με αυτά που είπατε εσείς. Πάντα είμαστε δεύτεροι μετά το στρατό, ε, μετά την Εκκλησία, συγγνώμη, όπως και εσείς. Και αυτό που μας παρουσιάσατε εδώ είναι μια σωστή αρχή. Πρώτα ξεκινάμε από τα νομικά και πολιτικά και νομικά θέματα και το νομικό πλαίσιο που το στείνουμε και μας επιτρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα να δω να πω δύο λόγια για τη σημασία της ε, μεταρρύθμισης του στρατού, γιατί θα είναι η αιχμή του δόρατος για τη μεταρρύθμιση ολόκληρης της σερβικής κοινωνίας. Πολιτικός πώς ε, θα έχει μεγάλη ορατότητα και μεγάλη σημασία και δεύτερον ε, έχει και την υποστήριξη του λαού. Και επίσης δίνει και κίνητρα στην υπόλοιπη κοινωνία να προχωρήσει με τι μεταρρυθμίσει. Αναφέρατε τις χώρες με τις οποίες έχετε σχέσεις. Η στατιωτική διπλωματία προχωράει χέρι-χέρι με την πραγματική δημοκρατία. Μπράβο σας. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει γνωστή η χώρα σας Χαιρετίζω επίση το γεγονό ότι σκοπεύετε να συμμετάσχετε και συμμετέχετε ήδη σε διάφορε πολυεθνικέ ε, επιχειρήσει και το γεγονό ότι ε, δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτό. Και το λέω αυτό γιατί από τη μία μέσα από τέτοιες επιχειρήσεις μαθαίνετε απίστευτα πράγματα, πολύ περισσότερα δεν πάνε να γίνουν 100 σεμινάρια. Είναι πολύ πιο σημαντικέ αυτέ οι επιχειρήσει, αυτά που μαθαίνετε, αυτά που αποκομίζετε από αυτέ τι επιχειρήσει επιτόπου. Επιπλέον, εν συνεχεία, δείχνετε στου συμμάχου σα ποιε είναι οι δυνατότητέ σα, ποιο είναι το δυναμικό σα. Ότι είσαστε αξιόπιστοι, αξιόπιστη δύναμη και νομίζω ότι αυτό αξιολογείται. Ας μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και ας μην πούμε ότι ε, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τη τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικές, ε, γιατί μπορεί να δοθούν μέσω αυτών και πολιτικές κατευθύνσεις. Κλείνοντας, το σύστημα στρατιωτικής ε, εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο γιατί πρέπει να ετοιμάσετε τους νέους που μπαίνουν στο στρατό με βάση το, το είδος του στρατού που θέλετε να οικοδομήσετε, αλλά και το τι του διδάσκεται. Όχι μόνο στρατιωτικό πώς αλλά και πολιτικό πώ. Προσπαθώντα να δημιουργηθεί μια νέα νοοτροπία για το σερβικό στρατό. Καλή επιτυχία λοιπόν. Και εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Merci, Ευχαριστώ κύριο Κούκαν, πρόεδρος ε, της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις Ευρώπης ε, Νοτιοανατολικής, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη. Ευρώπης. Καλωσορίζουμε τον Υπουργό Σουτάνοβατς. Σα ευχαριστώ που ήρθατε και μας δίνετε αυτές τις τελευταίες πληροφορίε για τις εξελίξεις στη χώρα σας στον τομέα του στρατού και της άμυνας. Θα αναφερθώ σε τρει τομεί τη σύντομη παρέμβασή μου. Καταρχά, η περιφερειακή συνεργασία. Όλοι τονίζουν τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας. Το μέλλον και τη μελλοντική συνεργασία των χωρών της περιοχής μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αυτό ισχύει και όλος ιδιαίτερος για τη στρατιωτική συνεργασία. Και από ό,τι είπατε, Υπουργέ, μια χαρά τα πάει η Σερβία. Αναφερθήκατε στις συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής και νομίζω ότι και η συνεργασία με την K4 είναι απτή. Σας ενθαρρύνω να προχωρήσετε έτσι και στο μέλλον για το ΝΑΤΟ. Από το 1999, όταν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ βομβάρδισαν την ε, Νέα Ιουγκοσλαβία, οι σχέσεις με μεταξύ Σερβίας και των συμμάχων πέρασαν μια δύσκολη περίοδο και μαλακά το, και ήπια το αναφέρω. Αλλά έτσι είχαν τα πράγματα εκείνη την εποχή. Περισσότερε χώρε. Ε, στην περιοχή προχώρησαν σχετικά γοργά και έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ. Αλλά το θέμα του κοσυφοπεδίου επιβράδυνε τον, την πορεία προς τον ΝΑΤΟ της Σερβίας. Πέρυσι έγιναν διάφορες αλλαγές, θετικές θα έλεγα, το 2006 η Σερβία ε, μπήκε στην εταιρική σχέση για την ειρήνη και πέρυσι συμφώνησε για το πρώτο πρόγραμμά τη με το ΝΑΤΟ. Ε, ετοιμάζει την πρώτη αποστολή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ η Σερβία και επίσης πολύ σημαντικό είναι η αντίληψη των συμμάχων για τη Σερβία. Βελτιώνεται και οι Σέρβοι πολιτικοί χρησιμοποιούν μια φρασιολογία, την φρασιολογία που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν λιγότερο συχνά. Και εσείς ο ίδιος αν χαρακτηρίσατε τη Σερβία πρόσφατα ως σύμμαχο, όχι ως εχθρό. Η Σερβία επίσης προοδεύει στη μεταρρύθμιση του στρατού για να στεφθεί από επιτυχία μας αυτή η προσπάθεια, οι εμπειρογνώμονες λένε ότι θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες από την κυβέρνηση. Σε επίπεδο στρατού και σε επίπεδο κυβέρνησης και Υπουργείου Άμυνας πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει ένα οργανωτικό δυναμικό, αλλά δυστυχώ δεν έχει εκμεταλλευτεί, ε, δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί απόλυτα ακόμα, δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα σε επίπεδο εφαρμογής λαμβάνοντα υπόψη τι ταραχές στο πολιτικό επίπεδο και την έλλειψη πολιτικής θέλησης και τα ανεπαρκή κονδύλια, αν θέλετε, για ορισμένες απαραίτητε μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, τα δύο θετικά στοιχεία που υπάρχουν θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Πρώτον, ένας επαγγελματικό στρατό. Ο κ. Σουτάνοβη είπε ότι μέχρι το τέλο του 2010 ο σερβικό στρατό θα σταματήσει την υποχρεωτική στατιωτική θητεία γενικού χαρακτήρα. Και ε, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της άμυνας, καθώς και η διεθνή συνεργασία για την ενδυνάμωση αυτού του κλάδου, που κατέστησε τον κλάδο αυτό το σημαντικό εξαγωγέα στην περιοχή, το σημαντικότερο εξαγωγέα στην περιοχή, βοήθησε την οικονομία της χώρας. Όλα αυτά είναι θετικά. Και έτσι θέλω να τελειώσω. Θέλω να ενθαρρύνω τον Πρωθυπουργό, τον ε, Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Σουτάνοβατ, να συνεχίσει αυτό το σημαντικό έργο, ε, σημαντικό για το μέλλον τη χώρα. και θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε την Σερβία στη μελλοντική της ευρωπαϊκή πορεία. Ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την νοτιοανατολική Ευρώπη, σας διαβεβαιώ ότι η δική μας αντιπροσωπεία κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τις χώρες στην περιοχή και τη Σερβία και θα συνεχίσουμε έτσι στο μέλλον. Καλή τύχη, κύριε Υπουργέ. Merci. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κατσίν που είναι και εισηγητής ε, για τη Σερβία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα σκοπό να μιλήσω σερβικά, αλλά δυστυχώς δεν είναι ακόμη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω όμως ότι η σημερινή επίσκεψή σας ε, θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη φιλοδοξία στην ε, Σερβία προκειμένου να φτάσουμε κάποτε ε, σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω γιατί μας παρουσιάσατε αυτό το πρόγραμμα μετάβαση, μετάβασης και ε, του σερβικού στρατού. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να μην ξεχνούμε ότι ένα από τα βασικά κριτήρια της δημοκρατίας είναι 100% πολιτικός έλεγχος ε, των στρατιωτικών δυνάμεων. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν έτσι τα πράγματα στη Σερβία. Μετά από κάποιες ε, αλλαγές ε, στο σύστημα μυστικών υπηρεσιών, κάποιοι άνθρωποι που δεν υπήρχαν εμφανίστηκαν και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό γιατί ο κύριος Κάρατζης είναι ήδη στη Χάγη είναι, εγώ είμαι σε μία μήχανη θέση γιατί είμαι εισηγητή για τη Σερβία, αλλά δεν υπήρχε έκθεση πέρσι για τη Σερβία. Ε, θα πρέπει να αρχίσουμε τη διαδικασία επικύρωσης ε, της μεταρρύθμισης των σερβικών ενόπλων δυνάμεων, ε, όμως δεν υπάρχει κανένα τρόπο ε, να συγκρίνουμε με οτιδήποτε, με στοιχεία του παρελθόντος. Θα ήθελα πάντω να σα ευχαριστήσω για τι προσπάθειε σα ε, εντός ε, των στρατιωτικών δυνάμεων. Θα ήθελα να σα ζητήσω να ολοκληρώσετε τι προσπάθειε σα για τον κύριο Μλάντιτ. και επίση θα ήθελα να ζητήσω για να μπορέσουν να, ε, να μπορέσει να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Όσον αφορά τώρα τη στρατιωτική θητεία, την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, είναι γεγονό ότι η μεταρρύθμιση σα θα δημιουργήσει θέσει απασχόληση σε μια περίοδο οικονομική κρίση. Ευχάριστο αυτό και επικοδομητικό και θα ήθελα να σας ε, ευχηθώ κάθε επιτυχία γιατί το να εφαρμοστεί αυτό θα είναι δύσκολο. Μπορεί να υπάρξουν απρόβλεπτα προβλήματα που θα πρέπει να τα υπερβείτε. Είναι ε, εύκολο να κάνει κανείς εξαγγελίες αλλά η εφαρμογή μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν ολοκληρώνοντας να πω το εξή ότι ο κύριος Μπράμετς ε, θέλει να ολοκληρώσει ε, την ε, διαδικασία στη Χάγη και εμείς το περιμένουμε αυτό εναγωνίως Παρακαλούμε λοιπόν να επισπευθεί όλη η διαδικασία, να κάνετε κι εσείς μία ακόμη προσπάθεια, μία επιπλέον προσπάθεια. Θα εκτιμηθεί όλος ιδιαίτερος. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Θα, έχουμε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό και θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι διαβάζετε τις εκθέσεις μας και χαίρομαι γι' αυτό και ιδίως ε, εξέρω τον κύριο Κούκαν για αυτά που είπε Όπως ε, είπα προηγουμένως, είμαι πρώην μέλος του Κοινοβουλίου. Παλιά ακούγα τη δική του άποψη του κυρίου Πάσκου, τώρα ακούω, τώρα ακούω αυτό στη δική μου. Εμείς έχουμε ε, αναβαθμίσει την στρατιωτική μας εκπαίδευση στο επίπεδο της πρώην Ιουκοσλαβίας. Έχουμε μία από τις καλύτερες στρατιωτικές ακαδημίες στην περιοχή και έχουμε αυτή τη στιγμή στη Σερβία 11 υψηλού Επίπεδο αξιωματικού που βρίσκονται σε αυτή τη σχολή και έχουμε και αξιωματικούς από την Αλγερία που είναι εκεί για τεχνική εκπαίδευση. Θα έχουμε από τη Γερμανία, από την Τουρκία, ήδη είχαμε από την ε, Ρωσία, από την Μακεδονία, τη Βοσνία, Ζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα περήφανοι γιατί μπορούμε να αναπτύξουμε τέτοιες σχέσεις μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων της περιοχής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι άνθρωποι που φορούν στολή κατανοούν οι μεν τους δε πολύ καλύτερα από ότι οι πολιτικοί τους καταλαβαίνουν. Όταν μιλάτε για την αρρωγή στην υπόλοιπη κοινωνία και τον εξοπλιστικό τομέα της βιομηχανίας, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη πρόοδο σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς στη Σερβία, ακριβώς στον τομέα της εξοπλιστικής βιομηχανίας. Το 1999 είχε ουσιαστικά εξολοθρευτεί αυτή η βιομηχανία από τους φοβατισμούς του ΝΑΤΟ, αλλά έχει ανακάμψει και ελπίζουμε εφέτος να έχουμε ένα ακόμα μεγάλο συμβόλαιο για ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ακόμα κατά τη δική μου θητεία, που είναι ένα μεγάλο ποσό για την μικρή Σερβία. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της μεταρρύθμισης, ξέρω ότι σε όλες τις χώρες είναι δύσκολο να προβεί κανεί σε μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά θα ήθελα να πω στη δική μας περίπτωση έχουμε 36.000 άτομα στο μισθολόγιο μας, έχουμε 50.000 κρατούμενους, έχουμε 38 ε, στρατηγούς, αλλά έχουμε και κάπου 750 συνταξιούχους στρατη, στρατηγούς. Έχουμε λοιπόν την κληρονομιά της δεκαετίας του 1990 η οποία βαραίνει ακόμα για μας. Και κάναμε πολλές προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση. Αναφερθήκατε επίσης και στο θέμα του επαγγελματικού στρατού Μιλήσαμε για τους άνδρες που εκπαιδεύονται στη στρατιωτική ακαδημία, αλλά έχουμε στην στρατιωτική μας ακαδημία και γυναίκες οι οποίες εκπαιδεύονται για στρατιωτικά καθήκοντα <clears throat> ως αξιωματικοί. Μιλήσαμε για το θέμα της συνεργασίας ή της σχέσης τουλάχιστον με τον ΝΑΤΟ και εκεί είναι βαριά η κληρονομιά του παρελθόντος. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να περάσουμε κάποιες δύσκολες ε, έχουμε να ξεπεράσουμε κάποιες δύσκολες εποχές για να έχουμε αυτή τη σχέση, αλλά θέλουμε να είμαστε πραγματικά εταίροι με το ΝΑΤΟ και προσπαθούμε να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Μετά από αυτά τα καλά λόγια που άκουσα από τον κύριο Κατσίν, θέλω να σας πω για την τελευταία συνάντηση που είχαμε στο Βελιγράδι, όταν με ρωτήσατε για τον πολιτικό και δημοκρατικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, προσπάθησα να σας πείσω τότε ότι έχουμε πλήρη δημοκρατικό και πολιτικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων στη Σερβία, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δεν ήταν τόσο εύκολο να επιτευχθεί. Κάτι που είναι εξάλλου σημαντικό για μας είναι ότι κανείς στην Σερβία και ούτε και το δικαστήριο της ε, Χάγης δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος κρύβεται στο έδαφος μας ακόμα και ο οποίος είναι υπόδικος. Όπως είπατε βρήκαμε κάποιους από αυτούς οι οποίοι το από το δικαστήριο της Χάγης, το ποινικό δικαστήριο την πρώην Ιουκοσλαβία, τώρα πρέπει να υπάρξει η πολιτική απόφαση για την τωρινή κυβέρνηση, για μένα, για όλους. Αυτό είναι μια διαδικασία που θέλουμε να την υποστηρίξουμε πλήρως. Σε πρακτικό επίπεδο, ξέρουν οι χώρες σας τι κάνουμε για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε όσο δυνατόν ταχύτερο αν μου πείτε να το κάνουμε αύριο αυτό, αν μπορούσαμε θα το είχαμε κάνει. Μην έχετε καμιά αμφιβολία για όλα αυτά. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς εξαρτώμαστε από την έκθεση του Serge Bramets, προχωρούμε όμως παράλληλα στις μεταρρυθμίσεις μας. Αν αυτή η έκθεση από τον κύριο Bramets είναι θετικού χαρακτήρα, θα πρέπει να επιτύχουμε τα πρότυπα τα οποία αναφέρει αυτή η έκθεση. Προσπαθούμε λοιπόν να επιτύχουμε όλα αυτά τα πρότυπα και να τα πραγματοποιήσουμε και στην πράξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεύτερος γύρος. Ο κύριος Τάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να μεταφραστούμε δεν μπορούν να μεταφραστούν τα σερβικά. Θέλω να σας ε, καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πω ότι είναι μια πολύ θετική η εντύπωση αυτή που μας δίνεται ότι είσαστε ένας πολιτικός ηγέτης και όχι ένας αξιωματικός. Είσαστε στην ίδια περίπου ηλικία με μένα. Παλιά ήταν δεδομένο σχεδόν ότι ένας υπουργός άμυνα θα ήταν αξιωματικό του στρατού. Είναι μεγάλη η πρόοδο στο ότι τώρα είναι φυσιολογικό να είναι πολιτικό ο Υπουργό Άμυνα στη Σερβία. Και αυτό αποτελεί μια πραγματική διασφάλιση ότι βρισκόμαστε από κοινού στο σωστή κατεύθυνση. Ω πολιτικό και ω μέλο τη κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Τσβέτσκοβιτ και συνεργάζεται και με τον πρόεδρο Τάντιτς θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον των ευρωπαϊστικών πολιτικών δυνάμεων στη Σερβία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας. <clears throat> Ποιε είναι οι κύριες επιτυχίες της τρέχουσας κυβέρνησης, ποιοι είναι οι στόχοι που ακόμα παραμένουν για να επιτευχθούν και ποιε είναι οι κύριες τάσεις που διατρέχουν αυτή την ευρωπαϊστικού χαρακτήρα ε, ομάδα που έχει την εξουσία στο, Βελιγράδι. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι πώς εκτιλήσεται η συνεργασία στα θέματα άμυνας με την γειτονική Μακεδονία. Είναι δυνατόν να, κάνουμε, να πράξουμε περισσότερα. Υπάρχουν σχέδια για τη βελτίωση αυτής της συνεργασίας ακόμα περισσότερο. Και το τρίτο και τελευταίο μου ερώτημα για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν ε, οικοτολογίες σε σχέση με τη νέα σας στρατιωτική βάση κοντά στην Νης και κοντά φυσικά στα σύνορα με το κοσκοπέδιο. Λένε ορισμένοι ότι οι Ρώσοι βρίσκονται πίσω από αυτή τη νέα στρατιωτική εγκατάσταση και είναι άλλος ο πραγματικός στρατός αυτής της βάσης. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε κάποια εξήγηση τι ακριβώς κάνει αυτή η στρατιωτική βάση και πώς λειτουργεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοπά. Uh, Ευχαριστώ. Είναι μια μεγάλη χαρά κύριε Υπουργέ να σας έχουμε εδώ ενώπιόν μας. Η Σερβία αλλάζει ραγδαία, αλλάζει πολύ έντονα και παρακολουθούμε τις προσπάθειές σας για να μεταρρυθμίσετε το στρατιωτικό κατεστημένο στην Σερβία και από αυτά που ακούσαμε από εσάς είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι και από αυτά τα οποία ξέρουμε και από άλλες πηγές μας. Χαροποιούν και οι προσπάθειές σας για καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γείτονες χώρες γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της Ευρώπης, της προσέγγισης για την Ευρώπη. Το ερώτημά μου αφορά το ΝΑΤΟ. Μετά από την τραυματική εμπειρία του 1999, ποια είναι η θέση της κυβέρνησής σας σε σχέση με την πλήρη ένταξη της χώρας σας στο ΝΑΤΟ. Μπορούμε να φανταστούμε κάποια στιγμή που η Σερβία θα θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Και ποια είναι η άποψη της κοινή γνώμης, ποια είναι τα συναισθήματα στην κοινή γνώμη σήμερα για το ΝΑΤΟ και εφόσον έχετε συμμετάσχει ήδη στην εταιρική σχέση για την ειρήνη, ποια είναι η άποψη του κόσμου σε σχέση με τη συμμετοχή της Σερβίας στο PFP, στην εταιρική σχέση για την ειρήνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την πρώτη παρουσίαση που κάνατε και από αυτά που είπε ο Αρνό Ντάουνσον, ο πρόεδρος μας, φαίνεται ότι είναι πολύ θετική η υποδοχή σας στην Επιτροπή μας αυτή. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κοινή ευαισθησία ανεξάρτητα από γεωγραφικές ή παραταξιακές ταυτότητες των βουλευτών σε αυτήν την Επιτροπή. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να συγχαρώ τον κύριο Υπουργό για τις πληροφορίες που μας έδωσε που ήταν τεκμηριωμένες, θετικές, εξαντλητικές σε σχέση με τη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων σε σχέση με τις εξελίξεις σε όλα τα πλαίσια και σε όλα τα στοιχεία στον στρατό της Σερβίας, ώστε να πάρει ένα επαγγελματικό χαρακτήρα, μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, να δημοκρατικοποιηθεί. Εγώ έρχομαι από μια χώρα που έχει ένα διαφορετικό σημείο εκκίνησης. Εγώ δεν προέρχομαι από την Ανατολική Ευρώπη όπου ίσχυε στο παρελθόν η επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης και οι οποίες χώρες αντιμετώπισαν τον ΝΑΤΟ σαν μια απελευθερωτική δύναμη. Εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου όχι μόνο η αριστερά και η δεξιά πολλές φορές βλέπουν τις ΗΠΑ σαν μια κυριαρχική δύναμη η οποία είναι αρνητική από αυτή την άποψη, κυριαρχία τη είναι αρνητική και το ΝΑΤΟ σαν κάτι το οποίο μπορεί να είναι ανεπιθύμητο. Αυτό άλλαξε όμως πριν από 25 χρόνια στην Ισπανία και άλλαξε προς τα θετικά. Το κόμμα μου με επικεφαλή στο Φέλιπε Γκονθάλε, έκανε ένα δημοψήφισμα για την παρουσία τη Ισπανία στο ΝΑΤΟ. Είναι το μόνο τέτοιο δημοψήφισμα που έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, ίσω και ποτέ. Και χάρη στο δημοψήφισμα αυτό, χάρη στον προσωπικό κύριο του Φέλιπε Κονσάλη, ουσιαστικά καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το δημοψήφισμα με μικρή διαφορά. Και από, και, από εκείνη τη στιγμή και επέκεινα, ήδη και πριν από το 82, γιατί το δημοψήφισμα έγινε το 1986, η πολιτική του να ενσωματώνουμε τις ένοπλες δυνάμεις στο σύστημα των ε, Ηνωμένων Εθνών και στις διαδικασίες ειρήνης και είχε σαν αποτέλεσμα οι Ισπανικές ένοπλες δυνάμεις οι οποίες είχαν μια φραγκική ιδεολογία στο παρελθόν και ακόμα και ενεπλάξαν σε απόπειρε πραξικοπημάτων κατά της σοσιαλιστικής κυβέρνησης τα, οι ένοπλες αυτές δυνάμεις μετεβλήθησαν σε δημοκρατικές, αποτελεσματικές, πιστές στην εξουσία με δημοκρατικό έλεγχο και αυτή είναι η πορεία η οποία έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα χωρίς καμία δυνατότητα υπαναχώρησης και αναστροφής αυτής της πορείας. Είναι γεγονός ότι η πορεία αυτή είναι πολύ σημαντική και υπάρχουν και κοινά στοιχεία. Όταν ακούω την παρέμβασή σας θυμάμαι πάρα πολλά από αυτά τα οποία ζήσαμε στην Ισπανία πριν από 25 περίπου χρόνια. Τις ε, θετικές αυτές ειρηνικές επαναστάσεις που έχουν γίνει στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις. Γι' αυτό κύριε Σιουτάνοβιτς θέλω να σας συγχαρώ και επαναλαμβάνω αν θέλετε το ερώτημα που κάναν άλλοι συνάδελφοι για την ε, μελλοντική σχέση που θα έχει η χώρα σας με τον ΝΑΤΟ. Και ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο δεν είναι ίσως απαραίτητο να το πω εδώ γιατί όλοι είναι πεπισμένοι περί αυτού, δημιουργήθηκε κάποια στιγμή στο παρελθόν ότι η στρατιωτική δύναμη και η πολιτική δύναμη είναι σημαντικές, αλλά πρέπει να υπόκειται στρατιωτική δύναμη στην πολιτική δύναμη. Στη δεκαετία του 80 είχε αναφερθεί το θέμα αυτό από ένα, ένας πολιτικός σε ένα σε μια συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική εξουσία και πολιτική εξουσία και η πολιτική εξουσία και η στρατιωτική εξουσία και η δικαστική εξουσία πρέπει να υπόκεινται στη λαϊκή θέληση, σε ένα δημοκρατικό έλεγχο. Λοιπόν, η Ισπανία ήταν από τι πρώτε χώρε που κατάφερε να ξεπεράσει αυτήν την ιδέα μια χωριστή στρατιωτική εξουσία και πολιτική εξουσία. Σα ευχαριστώ λοιπόν για τι πληροφορίε που μα δώσατε. Merci, Ευχαριστώ, κύριο Γκαλέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τουλάχιστον επί 10 χρόνια παρακολουθούμε την ε, Σερβία να ακολουθεί μια ευρωπαϊκή πορεία που την ε, οδηγεί σε έναν δρόμο σύγκλησης με την Ευρώπη. Ε, πολύ θετικό το ότι βρίσκεστε στο πνεύμα των πολιτών σας στη δεύτερη θέση μετά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Παρότι από ό,τι βλέπω παίρνετε και κάποια μη ορθόδοξα μέτρα με αυτό το πακέτο μέτρων που παρουσιάζεται. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το νομοθετικό πακέτο το οποίο μας εξηγήσατε. Σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις ένα πράγμα είναι η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο <laughs> και τελείως διαφορετικό η εφαρμογή στην πράξη αυτών των ε, νομοθετημάτων. Χρειάζεστε την ε, στήριξη των ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν τέτοια δημοκρατική εμπειρία. Και κάτι πιο συγκεκριμένο. Γνωρίζετε τον ε, διαμεσολαβητή στο στρατό ο οποίος ε, προστατεύει τους στρατιώτες από την αφαιρεσία κάποιων ε, ανωτέρων τους. Υπάρχει αυτή η φιγούρα του διαμεσολαβητή. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε ένα νέο στρατό, κάτι τέτοιο. Ε, και μάλιστα σε ένα στρατό που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και ένα ειδικά χαματισμένο παρελθόν. Η Σερβία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη στην Κωνσταντινούπολη υπέγραψαν στις 25 Απριλίου μια δήλωση για την ειρήνη στην ε, περιοχή. Είναι μια θετική δήλωση. Αλλά τι πρακτικές συνέπειες έχει αυτό για τη Σερβία. Για να ενδυναμώσουμε την ειρήνη στην νοτιοανατολική Ευρώπη χρειάζονται και άλλες χώρες. Γιατί υπογράψατε τόσο λίγες χώρες αυτή τη δήλωση. Θα έπρεπε αυτός ο κύκλος των ανθρώπων που υπογράφουμε είναι πολύ πιο ευρύς. Των χωρών που υπογράφουμε είναι πολύ πιο ευρύς. Κύριε Υπουργέ. Ε, ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που είστε μαζί μας ε, σήμερα στην Υπεροτροπή ε, Άμυνας και Ασφάλειας και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτά που είπατε, ειδικότερα για την βούληση της χώρας σας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα βήματα που κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ τα υποστηρίζω πλήρως και η ομάδα μου επίσης. Το θέμα της απελευθέρωσης ε, των θεωρήσεων είναι επίσης κάτι το οποίο ε, σε μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίξαμε. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Κάποιοι προλαλήσαντες ε, σας ρώτησαν και εκείνοι, επειδή εγώ είμαι μέλος μιας ουδέτερης χώρας που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αναρωτιέμαι η ιδέα του να προσχωρήσει κανείς στο ΝΑΤΟ πώς θα εκλειφθεί από την κοινή γνώμη της Σερβίας λόγω της ιστορίας που έχετε με τον ΝΑΤΟ και τα προβλήματα που υπήρξαν ε, με τον ΝΑΤΟ πριν από 10 χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς πώς κρίνετε την κατάσταση ως προς αυτό. Είπε ο κύριος Ντονζό ότι εγώ ήμουν ε, συγγήτρια για το κοσυφοπαίδιο ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεπώς δεν θα σας εκπλήξει το ότι έχω κάποιες ερωτήσεις ως προς αυτό. Ένα ερώτημα λοιπόν μας είπατε ότι θέλετε να διατηρήσετε την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας που συμπεριλαμβάνει το κοσυφοπαίδιο, αλλά είπατε επίσης ότι θέλετε, είστε αποφασισμένος να βελτιώσετε την περιφερειακή συνεργασία. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρί να αναγνωρίσετε το κοσυφοπαίδιο, αν και ελπίζω να υπάρξει πρόοδο ω προ αυτό ε, στο μέλλον. Είπατε ότι υπάρχει καλή συνεργασία με την K4, κάτι το οποίο επίση υποστηρίζω και επίση ε, επενέσατε και την ε, EULEX για την δουλειά τη. Είπατε εσείς ότι θα θέλατε να συμμετέχετε σε αποστολές ΕΠΑ στο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι που θα εκτιμούσα όλος ιδιαίτερο. Αλλά εάν η απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι αυτή που επιθυμείτε, και αν τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναγνωρίσουν το κοσυφοπαίδιο. Εγώ δεν ήμουν ε, μεταξύ αυτών που το υποστήριξαν αυτό σε μεγάλο βαθμό αλλά βλέπω ότι de facto είναι πλέον πραγματικότητα. Για να βελτιώσουμε λοιπόν τη συνεργασία και για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους και την εργασία που επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια αυτή νομίζω ότι θα βοηθούσε να υπάρχει μια κοινή θέση ως προς αυτό. Αλλά το ερώτημα μου κινείται περισσότερο προς την εξή κατεύθυνση. Αν θέλετε να συμμετέχετε σε αποστολές ΕΠΑ στο μέλλον, τι θα κάνετε, μπορείτε ας πούμε στρατιώτες από το Κωσυφοπέδιο να συμμετέχουν. Ε, θα συμφωνούσατε εσείς με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ερώτηση, κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω και τα δικά μου συγχαρητήρια και το καλώς ήρθατε προς τον ε, αξιότιμο κύριο Υπουργό. Ε, να προσθέσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου εκείνα των συναδέλφων μου για την πρόοδο που έχει επιτελέσει η Σερβία και στον κρίσιμο τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η ευρωπαϊκή πορεία και η προοπτική ε, της Σερβίας γίνεται όλο και πιο χειροπιαστή, καθώς επίσης και η προοπτική πιο ουσιαστικών σχέσεων ε, με τον ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, αναφυσβήτητα. Ξέρω και όλοι φανταζόμαστε πόση προσπάθεια χρειάστηκε από τις προοδευτικές, φιλοπρόοδες και φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις στη Σερβία, ώστε να, μεταβληθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα η αρνητική και επιφυλακτική ψυχολογία της ε, κοινή γνώμης της Σερβίας και του λαού της Σερβίας όσον αφορά τις σχέσεις του με τον ΝΑΤΟ. Και αυτό έχει επιτελεστεί γιατί κάποιοι υπεύθυνοι πολιτικοί ανέλαβαν αυτό το δύσκολο έργο. Και γι' αυτό κανείς θα πρέπει να σας συγχαρεί και πάλι. Η ερώτησή μου ε, αφορά κυρίως την ενεξελίξη, αναδιάρθρωση ε, και την μεταρρύθμιση των, ε, στον τομέα της άμυνας και των ενόπλων δυνάμεών σας. Η ερώτηση είναι η εξής. Έχετε διαμορφώσει στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης ένα δόγμα αμυντικής πολιτικής. Το έχετε επεξεργαστεί. Και αν ναι, στο πλαίσιο αυτού του δόγματος, ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι στόχοι ποια είναι η ανάλυση και η αντίληψη για την απειλή, third perception. Ε, και αυτό είναι σημαντικό, διότι πάνω σε αυτό χτίζεται ή και αν θέλετε η αντίληψη που έχετε για την απειλή και οι προτεραιότητες επηρεάζουν και την δομή και την οργάνωση και τη λειτουργία του αμυντικού συστήματος και των ενόπλων δυνάμεων μιας χώρας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Merci. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, λέει κύριο ε, Λοιπόν, σε τρία χρόνια υπογράψαμε 17 συμβάσεις για στρατιωτική συνεργασία, μεταξύ των οποίων και με την ε, ομόλογό μου της ε, Σλοβενίας, που είναι έφεδρο, εφεδριλοχαγός. Εγώ δεν είμαι όμως στο στρατό αξιωματικό στη χώρα μου. Με ρωτήσατε για, ποιες για το ποιες είναι οι κυρίες απειλές που αντιμετωπίζουμε. Εγώ μίλησα με τον, ε, με τον πρωθυπουργό σας τη Σλοβενία και έχω συναντήσει όλους τους πρωθυπουργούς ουσιαστικά από τη Βιέννη ως την Άγκυρα. Νομίζω ότι όλοι μας αντιμετωπίζουμε την ίδια απειλή σε όλη την περιοχή αυτή θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε απειλές που δεν προέρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα. Είναι απειλές που συνάπτονται με το οργανωμένο έγκλημα που έρχεται από όλες τις περιοχές του κόσμου και διατρέχει όλη την περιοχή μας. Η περιοχή μας είναι γνωστή ως, ήταν στο παρελθόν, ως δρόμος του μεταξιού. Τώρα είναι ο δρόμος του εγκλήματος, λαθρεμπορία γυναικών, λαθρεμπορία ναρκωτικών, όπλων Υπάρχει μεγάλη διασπορά ε, πολεμικών υλικών τα οποία κυκλοφορούν παρανόμως. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτές τις ενέργειες και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Με ρωτάτε επίσης τι είναι αυτά τα οποία απετέλεσαν τις επιτυχίες της κυβέρνησής μας για τα οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι. Νομίζω ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στην καταπολέμηση του, του οργανωμένου εγκλήματος. Πέρσι επιτύχαμε πολλά αντιμετωπίζουμε πολλούς ε, εγκληματίες και μέσα στο τελευταίο χρόνο περάσαμε ένα νέο νομοθέτημα με το οποίο έχουμε τη δυνατότητα κατάσχεσης των ε, προσόδων των οργανωμένων εγκληματι... εγκληματιών μάλλον και χθες ο Υπουργό Δικαιοσύνη μας είπε ότι μπορέσαμε να δημεύσουμε με τον τρόπο αυτό περίπου 100 εκατομ... Ε, αγαθά αξία ενό εκατομμυρίου ευρώ. Συνεργασία με τη Μακεδονία ή με την πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι πολύ καλή. Υπογράψαμε μια συμφωνία μαζί τους πέρσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μου ήταν πρόσφατα στο μοναστήρι στην Πίτολα όπου συναντήθηκε με τον ομολογό του εκεί. Έχουμε κάποιους αξιωματούχους οι οποίοι βοηθούν στην εκπαίδευση στην τοπική στρατιωτική ακαδημία και εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε τη συνεργασία μας με την ε, Μακεδονία. Θέλουμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε μαζί τους για να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο στρατιωτικής συλλογής πληροφοριών. Ξέρετε ότι είχαν προβλήματα σε ορισμένε επαρχίες τους με οργανωμένες ομάδες και τρομοκράτες. Η περιοχή των συνόρων της Σερβίας με την ε, Μακεδονία είναι πολύ κοντά στα σύνορα του πεδίου και γι' αυτό αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και τη συνεργασία όλων των, όλων των ε, χωρών αυτών για να επιληθεί το πρόβλημα. Επειδή τώρα μπορεί να υπάρχει κάποια παρεξήγηση αυτή η, η βάση που έδειξαν κοντά στον Πούνοβα και όχι στην ε, Νης είναι μια κανονική στρατιωτική βάση η οποία ξεκίνησε να οικοδομείται το 2003 για στρατιωτικούς στόχους και αστυνομικούς στόχους. Στη συνέχεια οι αστυνομικές δυνάμεις είπαν δεν θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν. Ο στόχος μας είναι να είναι μια φάση η οποία θα είναι διαλειτουργική για να μπορεί να υποστηρίξει και δραστηριότητες εκπαίδευσης για ειρηνευτικές ε, αποστολές. Ο στόχος μας είναι να μπορεί να υποδεχθεί και εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους από άλλες χώρες και από την άποψη αυτή η βάση θα μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολεί στη Σερβία. Όπως ξέρετε, είμαστε μέλη της εταιρικής σχέσης για την ειρήνη από το 2006, αλλά δεν έχουμε ακόμα ανοίξει ένα επίσημο γραφείο στην έδρα του ΝΑΤΟ. Η ιδέα μας είναι να το κάνουμε αυτό εφέτος και να φέρουμε σε πέρα στο σύνολο των δραστηριοτήτων για την ε, εταιρική σχέση με την ειρήνη, ότι κάποιοι που υποστηρίζουν το ΝΑΤΟ μου είπαν τι συνεργασία θέλουμε να έχουμε με το ΝΑΤΟ, εγώ είπα θα μπορούμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο της Αυστρίας ή της Σουηδίας, δηλαδή μέσα στα πλαίσια μιας κάποιας ουδετερότητας. Με ρωτάτε αν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε ειρηνευτικές ε, διαδικασίες, αν θα συνεργαστούμε με στρατιώτες από το Κοσφοπέδιο. Εγώ δεν ξέρω το Κοσφοπέδιο να έχει στρατό, αν έχετε κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το θέμα αυτό, ίσως θα είναι χρήσιμο να με πληροφορήσετε και εμένα. Φαντάζομαι ότι αυτό το ερώτημα αναφέρεται στο απότερο μέλλον. Για το κοσφοπέδιο ξέρετε ότι εμείς έχουμε δει μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Δεν υπήρξε καμία στρατιωτική δράση, καμία στρατιωτική επιχείρηση στο Κόσοβο και δεν εφαρμόσαμε καν εμπάργκο κατά του κοσμοπεδίο. Εμεί θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό με διαπραγματεύσει, με διπλωματικέ ενέργειε. Πιστεύω ότι είναι ο μόνο και ο καλύτερο τρόπο να λυθούν όλα τα προβλήματα τα οποία μπορεί να ανακύψουν στην περιοχή μα. Για τον διαμεσολαβητή στο στρατό, και αυτό ίσω είναι πάρα πολύ προχωρημένο για μας, ίσως πάρα πολύ σύγχρονο, αλλά υπάρχουν επιθεωρητές από που ελέγχουν το στρατό, υπάρχουν διάφορα επίπεδα εσωτερικού ελέγχου μέσα στο στρατό, από την στρατιωτική αστυνομία από, με, που προχωρούν προς τους ε, επιθεωρητές και τον επόμενο μήνα προβλέπουμε να δημιουργήσουμε μια γενική επιθεώρηση για τις υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών και κατασκοπίας και αντικατασκοπίας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν και το οποίο στο μέλλον θα πρέπει να είναι κάτι το δεδομένο για να είμαστε στο επίπεδο των χωρών, των προτύπων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό εγώ διαβάζω όλη την αλληλογραφία που έρχεται σε μένα από οποιοδήποτε και από τον τελευταίο κληρωτό. Όποιο μου στέλνει ένα γράμμα, το διαβάζω εγώ προσωπικά. Γι' αυτό δεν χρειάζομαι κάποιο διαμεσολαβητή. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, <clears throat> εγώ πάντα πληροφορούμε γι' αυτό. Βλέπω την αλληλογραφία που με περιμένει και είμαι έτοιμο να αντιμετωπίσω τα θέματα αυτά και δεν σταματάμε να εξετάζουμε αυτή την αλληλογραφία. Έχουμε διαμεσολαβητές στη Σερβική ε, στο σερβικό κράτος μπορούν όσοι θέλουν να προσφύγουν σε αυτόν αλλά ξεβλέπετε ότι δεν, είναι μια, δεν υπάρχει πια ταραχοποιό, ταραχοποιός χαρακτήρα στη Σερβία είμαστε πια τμήμα της λύσης των προβλημάτων και όχι της δημιουργίας των προβλημάτων <clears throat> για τη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Βοσνίας εγώ υπέγραψα μια συμφωνία συνεργασίας και με τη Βοσνία και με την Τουρκία έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τις δύο στρατιωτικές αυτές δυνάμεις Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία με τη Βοσνία, γιατί γνωρίζετε ποια ήταν η κατάσταση στο παρελθόν. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία μόλι πριν από δύο χρόνια και αυτή τη στιγμή έχουμε θαυμάσια συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνα τη Βοσνία και έχουμε ενθαρρύνει τον Βόσνιο Υπουργό να συμμετέχει η χώρα του σε ειρηνευτικέ ε, αποστολέ. Δεν ήταν πολύ εύκολο να το δεχτούν αυτό στη Βοσνία, αλλά επίση και με τι ε, τουρκικέ ενόπλε δυνάμει Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Είναι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν τους αξιωματικούς μας και από του χρόνου θα έχουμε ένα στρατιωτικό από την Τουρκία, ο οποίος θα βρίσκεται στη δική μας στρατιωτική ακαδημία. Αυτά λοιπόν για τη συνεργασία με τις χώρες αυτές. Δύο ακόμα παρεμβάσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που απαντήσατε και στις δικές μου ερωτήσεις. Ίσως δεν έπρεπε να είχα αναφέρει τους ε, στρατιώτες. Ε, τμήμα της ΕΠΑ είναι και πολίτες, όπως αστυνομικοί κτλ. Ε, εν πάση περιπτώσει, τώρα μιλάμε για το μέλλον, όχι για το τώρα. Είπατε επίσης ότι θέλετε να επιλύσετε τα προβλήματα και να βρείτε λύσεις, όχι στρατιωτικές, αλλά μέσω διαπραγματεύσεων. Ε, το υποστηρίζω πλήρως. Είναι σωστή προσέγγιση αυτή. Είπατε επίσης όμως ότι ότι η κυβέρνησή σας δεν έχει επιβάλει εμπάργκο στο κοσυφοπέδιο. Το ξέρω αυτό. Επίσης είπατε ότι είσαστε υπέρ της ε, περιφερειακής συνεργασίας, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει α, ε, εμπάργκο ε, για την ε, Σερβία και για την ε, και για το κοσφοπέδιο στα πλαίσια της ΕΖΕΣ. Σας ευχαριστώ που Αναφερθήκατε στην Αυστρία, σε χώρες ουδέτερε, ε, οι οποίες δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, αλλά που μπορούν σε κάποιες ε, να συνεργαστούν στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Ο κ. Κομουτσάκο, ε, να επανέλθω στην ερώτησή μου, κύριε Υπουργέ. Έχετε εκπονήσει ή είσαστε σε φάση εκπόνησης μιας, πλαισίου αμυντική πολιτικής και ποιε είναι οι προτεραιότητε αυτή τη στρατηγικής, της αν υπάρχει. Και ποιε είναι οι απειλέ που εκτιμάτε, ποια είναι η αξιολόγηση των απειλών ε, στα πλαίσια της στρατηγική σα. Ο Υπουργός. Για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Θα το διαβιβάσω στον Υπουργό Εμπορίου αυτό το ερώτημα για το εμπορικό εμπάργκο. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Όταν ήμουν μέλος του... Τώρα μάλλον που είμαι μέλος του Κοινοβουλίου βλέπω όλα τα προβλήματα και πώς συνδέονται μεταξύ τους. Τώρα αναφερθήκα σε στρατιωτικούς και ε, αστυνομικούς. Ε, για αυτό το πρόβλημα ε, θα το αφήσω όταν εμφανιστεί. Έχουμε τόσα προβλήματα να επιλύσουμε τώρα που δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Για την α, αμυντική πολιτική μας. Έχουμε μία πολιτική αμυντικής προστασίας και δεν θεωρώ ότι καμία χώρα γύρω από τη Σερβία συνιστά απειλή στρατιωτική απειλή. Δεν υπάρχουν τέτοιες απειλές μεταξύ των χωρών της περιοχής. Πρέπει να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε τις ασύμετρες διεθνείς απειλές για την περιοχή. Μπορώ να σας μοιράσω και αυτό το έγγραφο, το οποίο δεν είναι μυστικό και μπορείτε να ενημερωθείτε για το αμυντικό μας δόγμα. Ευχαριστώ και στα ελληνικά, λέει ο Υπουργός. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα κλείσουμε το πρώτο τμήμα αυτή τη συνεδρίασης. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις, αυτή την παρέμβαση του Υπουργού, να έχουμε μια άμεση ανταλλαγή απόψεων. Βλέπουμε απτές εντυπωσιακές προόδους που έχει κάνει η Σερβία. σε αυτό το τομέα ε, είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα που θιοθετήσετε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, μπορείτε να επανέλθετε στην ε, υποεπιτροπή μας και ούτως ή άλλως ε, πολύ σύντομα θα πάνε κάποια μέλη της Επιτροπής μας στη Σερβία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία μας. Θα κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. Ευχαριστώ.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

η να οφείλαμε σε αυτά η η τα συνδέσματα του υποβαθμισμένο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

Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να υποδεχτώ την κυρία Τζανέλα, που είναι τακτική θαμών της Επιτροπής μας. Έχουμε βέβαια πολύ φορτωμένη μέση σε δεν έχουμε τον χρόνο να τα εξετάσουμε όλα τα σημεία, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο ζητήματα για τα οποία θα ήθελα να μπορούμε να προχωρήσουμε σε συζήτηση. τα πυρηνικά του Ιράν μετά από την ε, επαφή που είχαμε με τον κύριο Μοτακίτ, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την πολύ καλή ε, ενημέρωση που μας έχετε εδώ στο παρελθόν για τα θέματα αυτά. Θα μπορούσα λοιπόν να σας παρακαλέσω να γυρίσουμε και πίσω στην, ε, στα ποινικά του Ιράν και τη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Βασιλείας και Ιράν, πώς αναλύεται από τεχνική έποψη αυτή την συμφωνία και επίσης να σταθούμε στην συνδιάσκεψη για τη μεταρρύθμιση της συνθήκης μη διασποράς των πυρικών όπλων που μόλις έχει υπερατωθεί και στην οποία συμμετάσχατε. Θα θέλα να έχω και τις απόψεις σας για τα πορίσματα αυτής της συνδιάσκεψης και τις επιτυχίες και αποτυχίες αυτής της συνδιάσκεψης. Θα χαιρόμουν πολύ να μπορέσετε να μας πείτε ποιες είναι οι απόψεις και να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα αυτά. Προηγουμένως <clears throat> στην Washington, είχε λάβει η χώρα η διάσκεψη για την ποινική ασφάλεια και πριν από την, συμφωνία της νέα, από την υπογραφή της νέας συμφωνίας START είχε προηγηθεί. Αυτά είναι θέματα λοιπόν τα οποία μας ενδιαφέρουν, αλλά θα σας αφήσω το λόγο για να αναφερθείτε σε αυτά τα θέματα. Πώς θέλετε να τα παρουσιάσω τα θέματα, να μιλήσω καταρχάς για το Ιράν. Μία ενημέρωση για το Ιράν. Δεν είχα τη δυνατότητα να παραστώ στη συνάντηση της Επιτροπής χθες με τον Ιρανό Υπουργό. Μπορώ λοιπόν να αναλύσω στην Επιτροπή σας την κοινή δήλωση μεταξύ Ιράν, Βραζιλίας και Τουρκίας. Όπως ξέρετε, μετά από την τελευταία συνεδρίαση μεταξύ του Χαβιέρ Σολάνα και του Ζαλίλη την 1η Οκτωβρίου στη Γενέβη. Ένα από τα σημεία του μνημονίου, της συμφωνίας που υπήρχαν μεταξύ του Ζαλίλη και του Σολάνα ήταν η συμφωνία επί της αρχής του Ιράν να εξάγει 1.200 κιλά ουρανίου ελαφρώς εμπλουτισμένου για να υπάρξει μια ανταλλαγή πυρηνικού καυσίμου για τον αντιδραστήρα της Τεχεράνης που κατασκευάζει ισότοπα. Είναι μια συμφωνία επί της αρχής, γιατί οι τεχνικές λεπτομέρειες θα έπρεπε να ολοκληρωθούν στην συνεδρίαση των Γενικών Διευθυντών της Παγκόσμιας, της Διεθνούς μάλλον Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας. Η συμφωνία αυτή είχε σαν σκοπό να λειτουργήσει Ω μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης στα πλαίσια μιας επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ των ομάδων των διαπραγματευτών ε, στην οποία ο Χαβιέρ Σοράνα ήταν εκπρόσωπος και του Ιράν. Επίσης, ξάγοντα 1.200 ε, κιλά ε, τον Οκτώβριο, αυτό ήταν το μεγαλύτερο τμήμα του ουρανίου που είχε παραχθεί στο Ιράν και που ήταν ελαφρώς εμπλουτισμένο. Ο σκοπός ήταν λοιπόν να κερδίσουμε χρόνο για τις διαπραγματεύσεις, να ηρεμήσουν τα πνεύματα της διεθνούς, στη διεθνή κοινότητα και να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτή η συμφωνία ολοκληρώθηκε σε μια συνεδρίαση στα μέσα Οκτωβρίου στη Βιέννη υπό την Προεδρία Παραντέη υπήρξε μια συμφωνία με την συμμετοχή της Γαλλίας, Γαλλίας, ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δύο-τρεις μέρες μετά η Γαλλία, η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείες επιβεβαίωσαν τη συμφωνία ε, για αυτή τη συμφωνία, για αυτό το deal, ενώ το Ιράν δεν επιβεβαίωσε την ε, συμφωνία του και επομένως είχαμε μια πλειάδα δηλώσεων στον τύπο επικριτικών, με διάφορες ε, μεταβλητές και παραμέτρους, αλλά ποτέ μια συμφωνία στο κείμενο της συμφωνίας, ποτέ δηλαδή το OK του Ιράν στο κείμενο της συμφωνίας της Βιέννης. Στο μεταξύ, το Ιράν αποφάσισε να ξεκινήσει τον εμπλουτισμό κατά 20%. Πέρασε από έναν εμπλουτισμό ε, κάτω από το 5% σε ένα εμπλουτισμό λίγο κάτω από το 20%. Υπό το πρόσχημα ότι θα πρέπει το ίδιο το Ιράν να παρασκευάζει τα καύσιμα για τον αντιδραστήρα του στην ε, κατάσταση ερευνητικού χαρακτήρα της Τεχεράνης. Φυσικά, ο εμπλουτισμός ε, μέχρι 20% είναι συνιστά μείζωνα ανησυχία. Γιατί όταν εμπλουτίζουμε μέχρι 20% τεχνικός πώς αυτό σημαίνει ότι είμαστε στα μισά του δρόμου που πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε σε μια στρατιωτική χρήση. Γιατί τεχνικός πώς για να περάσουμε από το 5% στο 20% απαιτεί τον ίδιο χρόνο και την ίδια προσπάθεια όπως το να περάσουμε από το 50 ας πούμε στο 90. Μια τεράστια προσπάθεια, δηλαδή 50 ως το 20, ε, μετά 20-50 κτλ. Όσο αυξάνει το ποσοστό εμπλουτισμού, ε, η προσπάθεια αυξάνει. Γι' αυτό λοιπόν το 20% μας ανησύχησε τα μάρλα. Το Ιράν δεν δέχτηκε τη συμφωνία του Οκτωβρίου και άρχισε να εμπλουτίζει μέχρι 20%. Σε αυτή τη συνεδρίαση τώρα με τους προέδρους, το, τον πρόεδρο μάλλον της Βραζιλίας και τον Τούρκο Υπουργό, συμφώνησαν σε μια κοινή δήλωση που περιλαμβάνει μια συμφωνία επί της αρχής του Ιράν να εξάγει προς την Τουρκία 1.200 κιλά ουρανίου αυτό το ουράνιο θα ελέγχεται, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ελέγχου που δεν είναι όμως πολύ συγκεκριμένες. Το κείμενο της δήλωσης λέει ότι η ατομική η υπηρεσία μάλλον ατομική ενέργειας μπορεί να στείλει επιθεωρητές. Μπορεί. Αλλά είναι κάτι το δυνητικό. Και δεν λέμε ποιε είναι οι προϋποθέσεις και ποιε είναι οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών της Διεθνούς υπηρεσία ατομική ενέργεια. Επίσης υπάρχει μια προθεσμία ενό έτου για την προμήθεια πυρηνικού καυσίμου. Κάτι που θεωρείται ανεπαρκές από αυτούς θα πρέπει να δώσουν αυτό το πυρηνικό καύσιμο. Και δεν υπάρχει καμία ένδειξη, αν ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, ότι το Ιράν θα είναι έτοιμο να σταματήσει τον εμπλουτισμό του Ιρανίου κατά 20%. Αυτό σημαίνει ότι το Ιράν... Α, να σας πω και κάτι άλλο. Στη δήλωση προς τον τύπο, οι θύνοντες του Ιράν επιβεβαίωσαν ότι θέλουν να συνεχίσουν τον εμπλουτισμό του Ιρανίου κατά 20%. Η δικαιολογία που δώσανε, ενώ θα λαμβάναν το πυρηνικό καύσιμο από άλλες χώρες, δεν υφίσταται, είναι αβάσιμη. Γιατί να συνεχιστεί αυτός ο εμπλουτισμός. Επομένως, αυτή η συμφωνία απλώς αυξάνει και πολλαπλασιάζει τις ανησυχίες μας. Ούτως ή άλλως παραμένουν ερωτηματικά γενικής φύσεως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και το Ιράν δεν κάνει τίποτα για να τις διασκεδάσει. Γιατί το επίπεδο συνεργασίας του με την Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας δεν βελτιώνεται. Ε, η παράγραφος 9 αυτής της δήλωσης λέει ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις, αλλά διευκρινίζει επί των κοινών σημείων της πρότασής. Αν κοιτάξετε την ε, Ιρανική πρόταση, η οποία έγινε πριν από ένα χρόνο, δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στο Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν δηλαδή είναι έτοιμο ε, για διαπραγματεύσεις και για συναντήσεις με τους έξι και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προβλήματα του περιβάλλοντος, της αλλαγής του κλίματος, τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, τη μείωση του, της στόχιας στον πλανήτη κτλ. Αλλά όχι για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και σας το λέω, γιατί εγώ συμμετείχα σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις από το 2004 και μετά. Όταν τους λέμε, δεν θα πρέπει να συζητήσουμε το πρόγραμμά σας. Λένε, το πυρηνικό μας πρόγραμμα δεν τίθεται ως ε, προσυζήτηση. Δεν είναι θέμα προσυζήτηση. Αυτή είναι η θέση τους. Να γιατί λοιπόν αυτή η κοινή δήλωση μεταξύ Ιράν, Βραζιλίας και Τουρκίας ε, θεωρούμε ότι θέτει πάρα πολύ, πολλά ερωτηματικά και πολλαπλασιάζει τις ανησυχίες. Καταλαβαίνουμε ότι το Ιράν χρησιμοποιεί αυτή τη δήλωση, ε, προσπαθεί τουλάχιστον, ότι φταίμε εμείς που η συμφωνία δεν οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο για να δείξει ότι αν οι συνομιλητές του είναι πιο λογικοί ή ήταν πιο λογικοί θα ήταν δυνατή η τελεσφόρηση της συμφωνίας. Και για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την υιοθέτηση ενός ψηφίσματος ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την άλλη βέβαια αυτή η κοινή δήλωση δεν έχει πολλά θετικά στοιχεία. Φυσικά, φαντάζομαι ότι ο Γενικό Διευθυντή τη Υπηρεσία Ατομική Ενέργεια θα μπορούσε να συγκαλέσει μια συνεδρίαση με τι εμπλεκόμενε χώρε ε, στο προηγούμενο σχέδιο συμφωνία και αυτή η συνεδρίαση θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει ενδεχομένω κάποια πράγματα, κάποιε παραμέτρου. Δεν αποκλείεται λοιπόν να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε αν αυτό το σχέδιο συμφωνίας είναι χρήσιμο. Υπό τον όρο βέβαια ότι οι προϋποθέσεις θα είναι αποδεκτές. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι αυτή η ανταλλαγή μεταξύ ουρανίου ελαφρώς ε, εμπλουτισμένου και πυρηνικού καυσίμου δεν είναι το πρόβλημα με το Ιράν. Το πρόβλημα με το Ιράν είναι το πυρηνικό τους πρόγραμμα, το οποίο έχει πτυχές που μπορεί, που μας ε, εμβάλλουν τη σκέψη ότι έχει μια στρατιωτική διάσταση. Πέρυσι. Οι συνομιλίες που έγιναν με, τους, με τα τρία άλλα μέρη είχαν σε σκοπό να δείξουν ότι ήταν δυνατόν το Ιράν να υποφεληθεί από τη συνεργασία στα πλαίσια ενός ε, καθαρά μη στρατιωτικού προγράμματος. Ήταν ε, μια προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά δεν ήταν η λύση στο Ιρανικό πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, ακόμα και αν φτάσουμε σε μια συμφωνία, σε, σε αυτό το deal, αν, αν τελεσφορήσει αυτό το deal της Βιέννης, παρόλα αυτά πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Ιράν για να διευκρινίσουμε τους πραγματικούς στόχους του προγραμματός τους. Ευχαριστώ. Προτείνω να περάσουμε στην συνθήκη μη διάζωσης και μετά να μιλήσουμε για το Ιράν. Αν δεν υπάρχουν ε, πολλές ερωτήσεις για το Ιράν, ε, αν θέλετε δύο-τρεις ερωτήσεις. Ε, ο κύριος Γκουαλχέρη, ο κύριος Κουμουτσάκος και ο κύριος Μπουτικόφερ. Πρώτα ο κύριος Μπουτικόφερ. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κυρία Τζανέλα για, για την παρουσίαση που μας κάνατε και τις σκέψεις που εκθέσατε. Εγώ θα ήθελα να θέσω τώρα κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επιτυχία ή την αποτυχία της προσπάθειας του Ιράν μέσω των διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας με την Τουρκία και την Βραζιλία να διασπάσει το μέτωπο των δυνάμεων κατά του Ιράν. Εσείς τονίσατε τα ασθενή σημεία αυτής της συμφωνίας. Θα ήθελα τώρα όμως εγώ, πέραν της ιστορίας που, της θέσης μάλλον που υπάρχει μέσα στην, ε, πέραν της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε και τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πόσο επιτυχής ήταν αυτός ο ελιγμός του Ιράν σε διεθνές επίπεδο και σε ποιο βαθμό επηρεάζει τη θέση που είχαν αναλάβει οι πέντε συν 1. Ευχαριστώ κύριο Κουρμουτσάκο. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Τζανέλα για την πολύ καλή και πλήρη ενημέρωση και τις απόψεις της. Ε, αναφερθήκατε, η ερώτηση μου είναι αναφερθήκατε σε ορισμένα κρίσιμα σημεία της τριμερούς συμφωνίας ε, Ιράν-Τουρκίας-Βραζιλίας, ορισμένα σημεία που χρειάζονται διευκρινήσεις ε, και ε, μεγαλύτερη πληροφόρηση. Αυτό είναι σημαντικό και θα ήθελα να ρωτήσω, ε, υπενθυμίζοντας βεβαίως κάτι που όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα, εάν η Επιτροπή είτε εδώ στις Βρυξέλλες, είτε με τον εκπρόσωπό της στην Άγκυρα, ε, ζήτησε από τις τουρκικές αρχές πληρέστερη ενημέρωση και διευκρινήσεις ακριβώς για αυτά τα σημεία που μόλις πριν λίγο μας αναφέρετε ότι χρειάζονται μεγαλύτερη ανάλυση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εάν η Επιτροπή έχει προβεί σε αυτές τις ενέργειες και στο αίτημα πληροφόρησης από τις τουρκικές αρχές ή αν δεν το έχει κάνει, αν προτίθεται να το κάνει. Και αν το έχει κάνει, αν σας απάντησαν, τι σας απάντησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci, Monsieur Γουαλτιέρη, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ε, πλήρη παρουσίαση της κατάστασης. Μιλήσατε για την αρχική συμφωνία για την πρόταση αρχική συμφωνία για τα 1.200 κιλά, ε, που είναι ένα μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη, έτσι το αναφέρατε. Αν δεν ε, σας παρεξήγησα, ένα από τα στοιχεία αυτού του confidence building ήταν να παρεμποδίσουμε έναν εμπλουτισμό ενός, ε, μιας ποσότητας ουρανίου επαρκούς που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή μιας βόμβας. Και επομένως, Μία από τα βασικά προβλήματα στη συμφωνία είναι ότι παρότι υπάρχουν αυτά τα 1200 κιλά, στο μεταξύ το Ιράν συνέχισε το πρόγραμμά του. Εγώ διάβασα μια πρόσφατη συμφωνία της ε, Επιτροπής ε, Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας που εκτιμούσε την ποσότητα του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει το Ιράν παρότι οι πληροφορίες δεν ήταν ακριβείς για το κατά πόσον χρειάζεται τόσος χρόνος για να κατασκευαστεί η βόμβα. Υπάρχει μια εκτίμηση για την ποσότητα του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει μέχρι τούδε το Ιράν. Αυτό είναι το συγκεκριμένο μου ερώτημα. Και έπειτα, Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στα πλαίσια μιας τακτικής, ας πούμε. Υπάρχει μια στρατηγική ε, για τον περαιτέρω εμπλουτισμό. Αυτά. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Η Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, απαντώντας τον κύριο Μπούτι Κόφερ, ή στο ερώτημά του καλύτερα, είναι σαφές ότι το Ιράν προσπαθεί να διχάσει τη διεθνή κοινότητα. Αυτό είναι ο στόχος του Ιράν με την κοινή αυτή δήλωση που έκανε την Βραζιλία και την Τουρκία. Και είναι τακτικές που χρησιμοποιεί συχνά το Ιράν από την αρχή της διαμάχης αυτής για τα πυρηνικά. Είναι σίγουρα, υπήρξαν σίγουρα επιτυχίες στο να δημιουργήσουν διχόνοια στην κοινή γνώμη και στη διεθνή κοινότητα. Μεταξύ άλλων, γιατί σε γενικές γραμμές υπάρχει μια παλιά διαφορά απόψεων μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών και των ε, βιομηχανικών χωρών σε ό,τι αφορά την ε, μεταφορά τεχνολογίας. Το Ιράν δεν είχε ποτέ δυσκολίες να πει σε άλλες χώρες στον αναπτυσσόμενο χώρο ότι στην πραγματικότητα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν είναι προβλήματα τα οποία ότι το πρόβλημα είναι μάλλον ότι οι μεγάλες δυνάμεις, οι δυτικές δυνάμεις θέλουν να εμποδίσουν το Ιράν από το να αποκτήσουν την σύγχρονη τεχνογνωσία για τα πυρηνικά. Αυτό είναι μια, ένα επιχείρημα το οποίο έχει απήχηση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επομένως δεν είναι δύσκολο να επιτύχει το Ιράν στο στόχο αυτό. Θα επανέλθω αργότερα στην διάσκεψη για την μη διασπορά των όπλων. Στη διάσκεψη αυτή η οποία μόλις περατώθηκε στις, ε, στη Νέα Υόρκη έχει προσφέρει μια πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών και ιδιαίτερα στη Βραζιλία πραγματικά χάρη και τις αραβικές χώρες ότι στην πραγματικότητα το Ιράν φέρεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ευθύς. Αυτό το οποίο πιστεύω λοιπόν είναι ότι αυτό που είναι στην Νέα Υόρκη και αυτό το οποίο θα συμβεί στο μέλλον θα μας βοηθήσει να καταδείξουμε ότι στην πραγματικότητα εμείς είμαστε ειλικρινείς όταν λέμε ότι οι ανησυχίες μας είναι μονάχα για μια πιθανή στρατιωτική διάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ότι δεν μας ενοχλεί η συνεργασία για ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας και επομένω το σύνολο θέμα έτυχε χειραγώγησης σε κάποιο βαθμό. Για την Τουρκία τώρα. Έχουμε επαφές με τις τουρκικές αρχές <clears throat> για, το, για την υποτιθέμενη αυτή συμφωνία. Αλλά νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με το Ιράν μέσω μιας τρίτης χώρας. Ήδη είναι δύσκολο να διαπραγματευτούμε με το Ιράν <clears throat> και αν διαπραγματευόμαστε μέσω μια άλλη χώρα, τα μηνύματα μπορούν να στρεβλώνται, να έχουμε σπασμένα τηλέφωνα, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση. Πρέπει να έχει κάνει άμεσε διαπραγματεύσει. λοιπόν. Αυτό είναι λοιπόν μια πτυχή που εγώ δεν το ανέφερα. Είναι παράξενο ότι υπήρξε μια πρόταση από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν και άλλες τρει χώρε. Γιατί τώρα η συμφωνία αυτή τη χάνει διαπραγμάτευση με χώρες που δεν ήταν στη Βιέννη τον Οκτώβριο. Εάν πρόκειται να γίνει κάποια συμφωνία στην πρόταση συμφωνία τον Οκτώβριο θα έπρεπε να τύχει διαπραγμάτευση στην ίδια ομάδα. Άμα γίνει μια συμφωνία σε μια άλλη ομάδα, αυτό δεν έχει νόημα. Αυτοί που διαπραγματευθήκανε με το Ιράν τώρα δεν γνωρίζανε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είχαν θεσπιστεί τότε και δεν γνωρίζανε ακριβώς τι είχε ελεγχθεί τι είχε αρνηθεί το Ιράν να δεχτεί στο παρελθόν. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε. Αλλά εν τέλει, και εδώ έτσι απαντώ, όχι μόνο στον κύριο Κουμουτσάκο, αλλά και στον κύριο Γκουαλτιέρη, τελικά, σε τελική ανάλυση, νομίζω ότι οι χώρες οι οποίες εμπλέκονται σε αυτή τη συμφωνία, και σας λέω ότι εμπλέκονται, αλλά δεν υπάρχει κατά την άποψή μου ακόμα μια απόφαση για τα θέματα αυτά. Θα προσκληθούν μάλλον από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να συζητήσουν και να διευκρινίσουν τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας και θα δούμε τότε αν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε επί τη βάση αυτής της πρότασης συμφωνίας. Η πρόθεσή μας τον Οκτώβριο ήταν να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να αποτελεί μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συγχρόνως να συμβάλλει στην βελτίωση της γενικής ατμόσφαιρας, του γενικού κλίματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ποσότητες, οι ποσότητες έχουν διπλασιαστεί από τον Οκτώβριο. Έχουμε 2.400 κιλά χαμηλού εμπλωτισμού ουρανίου. Και αυτό είναι το δεύτερο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Γιατί δέχεται το Ιράν τη σημερινή συμφωνία και όχι τη συμφωνία του Οκτωβρίου. Γιατί ακόμα κι αν <clears throat> εξαγάγουν 1200 κιλά χαμηλού εμπλωτισμού ουρανίου, έχουν άλλα 1200 που έχουν μείνει τώρα στο Ιράν. Για, τον, για την εκτίμηση τη ποσότητα του εμπλωτισμένου ουρανίου στο Ιράνιο, εγώ μπορώ να πω μονάχα αυτό το οποίο λέει η Διεθνή Υπηρεσία ατομικής ενέργειας λέει 2.400 κιλά χαμηλού εμπλουτισμού. Αυτό είναι λοιπόν μια εκτίμηση που γίνεται από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας επί τη βάση του, των γνωστών εγκαταστάσεων εμπλουτισμού που είναι γνωστές στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα όμως για άλλους, ε, άλλες άλλες εγκαταστάσεις. Η εγκατάσταση του ΚΟΥΜ δεν είχε δηλωθεί στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Μόνο έγινε αυτό όταν το Ιράν κατάλαβε ότι όλοι ξέραν και τότε την έκανε γνωστή. Επομένως, δεν ξέρουμε αν μόνο αυτό το ουράνιο είναι στα χέρια του Ιράν. Και εδώ η δυσκολία είναι ότι όλοι μας έχουμε αμφιβολίες για το χρόνο που χρειάζεται το Ιράν για να παραγάγει πυρηνικά όπλα. Αν είναι οι μονάχα οι ποσότητε που ξέρουμε που έχει στη διάθεσή του το Ιράν, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, τουλάχιστον ένα χρόνο, ένα χρόνο μπορεί και περισσότερο χρόνο για να πετύχει να φτάσει σε ποιότητα οπλικού συστήματο. Χρειαζόμαστε περισσότερο ουράνιο, το φτάσουμε σε ε, εμπλουτισμό 90% να το μετατρέψει το ουράνιο σε όπλο, να έχει ένα βαλιστικό πύραυλο, ένα τρόπο να μεταφέρει, να εκτοξεύσει αυτό το όπλο το Ιράν, που αυτή τη στιγμή δεν το έχει. Όλα αυτά λοιπόν για να μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα χρήση πυρηνικών όπλων. Αλλά ίσως και για τη δημιουργία πυρηνικών όπλων πριν από 2-3 χρόνια είχε βρει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάποια σχέδια και σκαρυφήματα που έδειχναν ότι το Ιράν ξεκινούσε την παραγωγή όπλων. Ίσως υπάρχουν λοιπόν μελέτες για μετατροπή του ουρανίου σε πυρηνική κεφαλή, κάποιες ε, δοκιμές σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να κάνουμε μια εκτίμηση. Κύριε Πρόεδρε, Λίγο πολύ σύντομα θα ήθελα να πω. Καταλαβαίνω και λαμβάνω σοβαρά υπόψη αυτό που είπατε για τον κίνδυνο ε, του να εμπλακεί κανείς έμεσα σε διαπραγματεύσεις με τον Ιράν και μιλάω για την Τουρκία. Αλλά ίσως θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη επίσης ότι είναι μια υποψήφια χώρα η Τουρκία και τουλάχιστον θεσμικός ε, δεν θα έπρεπε να παρεκκλίνει από την ε, κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι ουσιαστικό θέμα αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να ζητήσουμε από τους Τούρκους να διευκρινίσουν ε, περισσότερο τη συμφωνία με το Ιράν. Θα πρέ... Λαμβάνω βέβαια πολύ σοβαρά υπόψη αυτό που είπατε για τις έμεσες συζητήσεις με την Τεχεράνη. Ευχαριστώ πολύ, το σημειώνουμε. Να συνεχίσουμε τώρα με τη δεύτερη πτυχή που αφορά την ενδιάμεση ε, αναθεώρηση της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η διάσκεψη αναθεώρησης για την μη διάδοση πυρηνικών όπλων ε, που έγινε στην Νέα Υόρκη το Μάιο ήταν επιτυχής. Και λόγω των εγγράφων που εγκρίθηκαν από τη διάσκεψη, αλλά και λόγω της συμβολής της ε, στην βελτίωση της σχέσης ε, μεταξύ των δυτικών και των αναπτυσσομένων χωρών. Βελτίωση που ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει. Το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε, το διαπιστώσαμε κατά τις τελευταίες μέρες, η αντίδραση του Ισραήλ ε, για την ε, συμφωνία που απετεύχθη για ε, την Μέση Ανατολή και θα αναφερθώ κάποια στιγμή αργότερα στην παρουσίασή μου για το θέμα αυτό. Το τελικό έγγραφο της διάσκεψης αναθεώρησης έχει δύο τμήματα. Υποθέτω ότι έχετε λάβει τα τελικά αντίτυπα. Το πρώτο τμήμα αφορά την αναθεώρηση, δηλαδή την εξέταση του πώς έχουν εφαρμοστεί τα άρθρα της συνθήκης, δυσκολίες, προβλήματα κλπ. Το τμήμα της αναθεώρησης είναι προϊόν ε, μιας ε, συλλογής ε, σχεδίων εκθέσεων ε, των προέδρων των διαφόρων επιτροπών που έχει ιδρύσει η διάσκεψη για την αναθεώρηση. Αλλά αυτά τα σχέδια εκθέσεων δεν εγκρίθηκαν από τα κράτη. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος στο τέλος της διάσκεψης για να, εξετάσουμε, για να εξεταστούν οι εκθέσεις αυτές. Δεν υπήρξε δηλαδή επίσημη διαδικασία έγκρισης. Είναι λοιπόν υπευθύνη του των προέδρων, αλλά σε γενικέ γραμμέ ε, αντικατοπτρίζουν ε, την ουσία των συζητήσεων στι διάφορε επιτροπέ. Το δεύτερο τμήμα αφορά το μέλλον και συμπεριλαμβάνει σχέδια δράσεων ε, για, τις ε, τρεις πυλώ, για τους τρεις πυλώνες, ε, τις ειρηνικές χρήσεις, την ε, μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Το δεύτερο τμήμα εγκρίθηκε ε, από την ε, διάσκεψη αναθεώρησης. Σας μίλησα για τα σχέδια δράσης. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα βήματα που τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να εφαρμόσουν. Για τον αφοπλισμό, Μιλούμε για 22 δράσεις και θα δείτε ότι η γλώσσα αυτού του τμήματος που έχει να κάνει με τον αφοπλισμό είναι πάρα πολύ έντονη. Αναφέρεται συγκεκριμένα στα πυρηνικά όπλα και λέει ότι τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευθεί, δηλαδή η γλώσσα είναι συχνά ε, τέτοια που δηλώνει νομική υποχρέωση. Υπάρχει επίσης η αρχή της ε, μη ανατρεψιμότητας, της διαφάνειας ε, ε, και της εφαρμογής των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της συνθήκης, ανάληψη υποχρέωσης κατάργησης των πυρηνικών όπλων, όπως επίσης και επίσπευσης συγκεκριμένη προόδου με σκοπό τον πυρηνικό αφοπλισμό. Και ειδικότερα η ειδικότερη αναφορά γίνεται στην επίσπευση της σταδιακής μείωσης της χρήσης όλων των πυρηνικών όπλων. Υπάρχει επίσης ειδική μνήμα όταν μιλάμε για πυρηνικά όπλα. Αυτό σημαίνει κάθε είδους όπλο σε κάθε ε, σε οποιοδήποτε μέρος και σε τακτικά όπλα που μπορεί να βρίσκονται κάπου αποθηκευμένα στην ε, Ευρώπη. Επίσης, ειδική μνήμα στην ε, σταδιακή μείωση του ρόλου των πυρηνικών όπλων στα στρατιωτικά δόγματα. Επίσης, έκκληση για περαιτέρω μείωση των, ε, του επιχειρησιακού καθεστώτος των ε, πυρηνικών όπλων, όπως επίσης ε, και την ενίσχυση της αμοιβαία εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Όσον αφορά τώρα την συνθήκη πλήρους απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών, δυστυχώς ισχύει μόνο για χώρες που ήδη έχουν προσχωρήσει στην συνθήκη αυτή και θα σας εξηγήσω γιατί. Επίσης, Όσον αφορά το σχάσιμο υλικό, αναφέρεται μεν, αλλά δεν ε, αναφέρεται τίποτε για το μορατόριουμ για το σκάσιμο υλικό. Η Κίνα προσφάτως υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια ως προς ε, την ε, χρήση πιο ε, ήπιας γλώσσας για, την, για τα θέματα σκάσιμου υλικού. Όπως είπα, οι περισσότερες δράσεις έχουν, αναφέρονται με πολύ έντονη γλώσσα και θα ήθελα να πω ότι για πρώτη φορά στο κεφάλαιο αυτό η γλώσσα ε, που χρησιμοποιείται αναφέρεται στο reporting ε, των κρατών μελών ε, στο μέλλον. Είναι πρώτη φορά που τα κράτη-μέλη δέχονται τέτοιου είδους αναφορά, γιατί μέχρι τώρα υπέβαλαν εθελοντικώς πληροφορίες. Βέβαια, αυτό δεν είναι αναγκαία κακό, Γιατί, για παράδειγμα, οι εθελοντικέ πληροφορίε που μα υπέβαλε φέτο η Γαλλία ήταν πάρα πολύ πλήρε. Αλλά τώρα πλέον υπάρχει μια υποχρέωση υποβολή εκθέσεων. Μετά υπάρχει ένα τμήμα που αφορά τη μη διάδοση με 24 ε, δράσει. Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές αυτό το κεφάλαιο για την μη διάδοση είναι λιγότερο φιλόδοξο και περιλαμβάνει λιγότερες υποχρεώσεις σε σχέση με τον αφοπλισμό. Σε περισσότερες περιπτώσεις αντί για ανάληψη δέσμευσης δέσμευση ε, η υποχρέωση, ε, ε. η ομάδα ΝΑΜ ήταν πάντοτε αλλεργική στο επιπρόσθετο πρωτόκολλο και στον έλεγχο των εξαγωγών, γιατί θεωρούν ότι αυτός είναι ένας τρόπος ε, παρακόλλησης της ε, ε, μεταφοράς τεχνολογίας και αυτή τη φορά έχουμε μια αρκετά καλή γλώσσα όσον αφορά τα, την, το επιπλέον πρωτόκολλο. Λέει ας πούμε ενθαρρύνει την σύναψη και την εφαρμογή επιπρόσθετων πρωτοκόλων το συντομότερο δυνατόν. Εφαρμογή μάλιστα προσωρινή μέχρι την έναρξη ισχύω του πρωτοκόλου. Άρα λοιπόν αναγνωρίζεται ο κανόνας ε, του ελέγχου των εξαγωγών όπως επίσης και των κατευθυντηρίων γραμμών ε, ε, στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού. Αυτό που είναι μάλλον αδύναμο είναι το τμήμα της ε, συμμόρφωσης. Ε, πολύ γενική γλώσσα, δεν ε, υπάρχει αναφορά στο Ιράν, δεν υπάρχει αναφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ε, μόνο για τον εσωτερικό κανονισμό της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και επίσης περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ε, και παραπομπής στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ε, Επίση, ε, υπάρχει ένα τρίτο κεφάλαιο με 18 δράσεις. Ε, πολύ επικοδομητική γλώσσα χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Κάπως μεγαλύτερο άνοιγμα, πιο πολυμερής προσέγγιση, αλλά Είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν ήταν πάρα πολύ δημοφιλέ το, αυτή η πολυμερή προσέγγιση. Υπάρχει επίσης ε, αναφορά στην πυρηνική ασφάλεια, όχι ειδική μνήμα στη Σύνοδο τη Ουάσιγκτον, αλλά ε, αναφέρεται σαφώς στην πυρηνική ασφάλεια και στην ανάγκη συμμόρφωσης ε, με τις σχετικές συμβάσεις για την ε, προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ε, την καταστολή δραστηριοτήτων πυρηνικής τρομοκρατίας ε, κλπ. Υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά τη Μέση Ανατολή. Το 1995 στην τότε διάσκεψη αναθεώρησης αποφασίστηκε μία εσαΐ επέκταση της συνθήκης, κάτι το οποίο όμως το φίλουμε ε, στην παράλληλη έγκριση ενός ψηφίσματος ε, για την Μέση Ανατολή και ζητούσε, το οποίο ζητούσε μία διπλή ελεύθερη ζώνη ελεύθερη ε, από πυρηνικά ζώνη στη Μέση Ανατολή. Η Αίγυπτος εκ μέρους της αραβικής ομάδας εδώ και μερικά χρόνια κατέστησε απολύτως σαφές ότι η διάσκεψη θα μπορούσε να είναι επιτυχής αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για κάποια βήματα για την εφαρμογή του ψηφίσματος για τη Μέση Ανατολή. Και έχουμε αποφασίσει, έχουμε καταλήξει σε ένα κείμενο που προβλέπει μία διάσκεψη που θα συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ε, η και από τις Ηνωμένε Πολιτείε, τη Ρωσία και το ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Διορισμός ενός συντονιστή και επιπλέον επιπρόσθετα βήματα όπως για παράδειγμα οργάνωση σεμιναρίων ε, για το θέμα αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο έχουμε οργανώσει και στο παρελθόν πριν από τη διάσκεψη ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι αρχέ αρχές ε, του 2011. Γίνεται αναφορά στο Ισραήλ στο κείμενο αυτό που αφορά τη Μέση Ανατολή, όμως δεν είναι στο διατακτικό του κειμένου, είναι στο προήμιο και λέει ότι η διάσκεψη αναγνωρίζει την σημασία της προσχώρησης του Ισραήλ ε, στην συνθήκη, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει ε, δεν αναφέρεται με αρνητικό τρόπο, απλώς αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αναφέρεται μάλιστα και στον Νετανιάχου και στο τι είχε πει ότι δεν θεωρείται ότι δεσμεύεται από την απόφαση που έλαβε ε, η διάσκεψη ε, μιας συνθήκης στην οποία δεν έχει προσχωρήσει το Ισραήλ. Μία από τις προκλήσεις λοιπόν που έχουμε να ε, αντιμετωπίσουμε είναι ότι πρέπει να δουλέψει όλο αυτό. Ήδη εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμαζόμαστε για το σεμινάριο αυτό. Πρέπει να προσεγγίσουμε το Ισραήλ και πρέπει να το πείσουμε τουλάχιστον να συμμετέχει σε ένα διάλογο για μια ζώνη ελεύθερη από πυρηνικά στην περιοχή και να τους πείσουμε ότι είναι και προς το δικό του συμφέρον. Αυτό είναι το μεγάλη πρόκληση που έχουμε, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δύο-τρία πράγματα τώρα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει, θα έλεγα, ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια αυτής της διάσκεψης. Ξέρετε ότι η Κάθριν έχει παρουσιάσει, έχει κάνει την ενακτήρια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση την πρώτη μέρα της συνδιάσκεψης και δόθηκε αυτή η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι δεν το επέτρεπαν απόλυτα οι κανόνες διαδικασίες αλλά ήταν αρκετά φιλελεύθερος ο πρόεδρος για να εξασφαλίσει τη συμφωνία των εμπλεκομένων ομάδων ώστε να γίνει αυτό το πράγμα. Η Προεδρία και εγώ υπήρξαμε πολύ ενεργοί στην, ε, στις διάφορες ομάδες εργασίας και ιδίως στην ομάδα που διαπραγματεύτηκε το σχέδιο δράσης την τελευταία μέρα της συνδιάσκεψης. Νομίζω ότι υπάρχει γενική συμφωνία όλων τώρα ότι ότι τα συμπράσματα της συνδιάσκεψης ήταν πολύ θετικά και επικοδομητικά. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθεαυτή και όχι ως Γαλλία, Αγγλία ή οτιδήποτε τέτοιο συμμετέχει στους τελευταίους γύρους των διαπραγματεύσεων. Για πρώτη φορά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ότι είναι ένα σημαντικό παίκτη στον τομέα τη μη διάδοση των ποινικών όπλων. Και σταματώ εδώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο, για την πλήρη αυτή παρουσίαση. Η κυρία Κόπα θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σα. Το ερώτημά μου αφορά το σεμινάριο για τη Μέση Ανατολή στο οποίο αναφέρθηκατε. Ίσως είμαι αφελής δεδομένης της θέσης του Ισραήλ και της θέσης του Ιράν. Τι ακριβώς περιμένετε να προκύψει από αυτό το σεμινάριο. Ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις αυτών των δύο χωρών. Δεν υπάρχει καμία θέληση από την Ισραηλινή κυβέρνηση να πράξει οτιδήποτε θα μπορούσε κανεί να ζητήσει από αυτούς ε, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Ακόμα και η αναφορά στο Ισραήλ στο κείμενο τους δυσαρέστησε Ξέρουμε και τη θέση της Ιρανικής κυβέρνησης. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν αυτού του σεμιναρίου. Απλώς να κάνουμε ένα σεμινάριο για τη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ερώτημά μου λοιπόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλα. Σας ευχαριστώ. Αναφέρατε πριν από λίγο ότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα συμμετέχει σε μια τέτοια διασκέψη και όχι μονο μόνο κράτη-μέλη της. Μέσα στα πλαίσια της ε, συνδιάσκεψης αυτής υπήρξαν κάποιες ε, αναφορές στα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με ένταση μεταξύ των πυρηνικών, των κρατών με πυρηνική ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών χωρίς πυρηνική ικανότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπήρξε κάποια τέτοια ένταση μέσα στις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο ερώτημα. Είπατε στην τελευταία σας ε, επισκέψη στην ε, υποεπιτροπή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πλήρες μέλος στην πρωτοβουλία για τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων αυτή τη στιγμή και ποια είναι η προσθέμενη αξία η οποία θα προκύψει για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν πράγματι γίνεται εκτή μέλος σε αυτή την πρωτοβουλία. Ο κύριος Μπουτικόφερ. <coughs> Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Μπουτικόφερ. μικρόφωνος. Σας ευχαριστώ για την εκτενή σας έκθεση. Αλλά Πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ απόλυτα με την κρίση που έχετε εκφέρει για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της συνδιάσκεψης για, για τη διασπορά των πυρηνικών όπλων, τη μη διασπορά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κεντρικού χαρακτήρα, έχει αποδυναμωθεί παράλληλα από το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για ένα συγκεκριμένο έγγραφο που να καλύπτει τα τακτικού χαρακτήρα πυρηνικά όπλα. Πιστεύω πράγματι ότι το τελικό αποτέλεσμα της διάσκεψης για τα τακτικά πυρηνικά όπλα είναι πιο ισχνό αυτή τη φορά, πιο ασθενές από ότι στην δήλωση της ε, συνδιάσκεψης αναθεώρησης του 2000 δεν πρέπει λοιπόν να αυταπατώμεθα. Υπάρχει ακόμα μια διαμάχη για τα θέματα αυτά και η χώρα μου, ιδίως η Γερμανία, είναι πολύ δυσαρεστημένη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κοινή στάση και ένα κοινό έγγραφο θέσης. Αυτό είναι τα παραδείγματα λοιπόν μιας αστοχίας του συστήματος του λεγόμενου γάλλο-γερμανικού άξονα. Τώρα, αν αντιμετωπίσω σε ευρύτερο πλαίσιο τα αποτελέσματα της συνδιάσκεψης, προφανώς υποστηρίζω την άποψή σας ότι υπήρξε κάποια σημαντική πρόοδος, ιδίως σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή. Αυτό ήταν πολύ χρήσιμο. Και επίσης το γεγονός ότι στη σελίδα 11 συμπεριλήφθηκε ένα κομμάτι κειμένου το οποίο αναφέρει ότι μια πλειοψηφία των χωρών οι οποίε είχαν εμπλακεί στι διαπραγματεύσεις θα θέλανε να υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τον αφοπλισμό των πυρηνικών δυνάμεων και αυτό ήταν ένα θετικό βήμα για μένα. Βλέπω όμως να υπάρχουν και αδυναμίες και αρνητικά αποτελέσματα στα πορίσματα αυτά. Και θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να μας δώσετε μια πιο ισορροπημένη εικόνα. <clears throat> Παραδείγματος χάρη όταν πρόκειται για τις ε, ευθύνες των κρατών με πυρηνική ικανότητα να σεβαστούν τις υπάρχουσες υποχρεώσεις που έχουν συνάψει σε σχέση με τα θέματα ασφαλείας, αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο συμφωνήθηκε. Δεν υπήρξε η δέσμευση, όπως το έπραξαν οι Κινέζοι, να υπάρξει δηλαδή μια δέσμευση, όπως έκανε οι Κινέζοι, να μην χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα εναντίον κρατών που δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βρίσκω λυπηρό εγώ. Και επίσης, σε σχέση με την αναγκαιότητα να υπάρχει μια συμφωνία για ανώτατο όριο στις ποσότητες χασίμου υλικού που έχει κάθε χώρα στη διάθεσή της και πάλι το τελικό κείμενο αναφέρεται στην διάσκεψη των ΗΠΑ για, την, ε, για τον αφοπλισμό ενώ η προηγούμενη μορφή του κειμένου θα είχε επιτρέψει να υπάρχει μια παραπομπή στην Γενική Συνέλευση των ΟΕΕ και θα είχε προτείνει να έρθει το θέμα αυτό στην 60η Σύνοδο του, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ως ένα φόρουμ για να προωθηθεί αυτό το θέμα, αν κάποια κράτη-μέλη του ΟΗΕ εξακολουθήσουν να μπλοκάρουν την πρόοδο στον τομέα αυτό. Είναι λοιπόν ισχνό το αποτέλεσμα. Δεν επιτέχθη αυτός ο στόχος που προανέφερα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες διασφάλισης και τα πρόσθετα πρωτόκολλα, είναι αποδυναμωμένη η φρασιολογία, η διατύπωση. Αναφέρονται τα εργαλεία αυτά σαν κάποια από τα στοιχεία της συμφωνίας, ενώ θα πρέπει να αναφέρονται ως κεντρικά, ως κομβικά στοιχεία και πιστεύω ότι θα έπρεπε να θεωρείται ως προϋπόθεση για την μεταλαμπάδευση τε, πυρηνικής τεχνολογίας το να είναι οι χώρες προς τις οποίες πηγαίνει η τεχνολογία μέλη της συμφωνίας αυτής. Επίσης, εσείς αναφέρατε το θέμα το, της παροχής αναφορών ως θετικό στοιχείο, ενώ προβλεπόταν η, η παρουσίαση αναφορών από τα κράτη-μέλη εκθέσεων ε, σε πολύ πιο έγκαιρο επίπεδο προβλεπόταν στην αρχή από ό,τι είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θέλω τώρα να συνεχίσω να αναφέρω όλα αυτά, αλλά ίσω θα πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι στι παρουσιάσει. Να μην λέμε μοναχά ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα, αλλά να φέρουμε και την αρνητική πλευρά. Και εδώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο είναι για μένα το πιο λυπηρό είναι ότι εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευκαιρία να προωθεί στη δική της ατζέντα για τα τακτικά όπλα πυρηνικού χαρακτήρα δεν κατάφερε να το κάνει στην πραγματικότητα. Ο κύριος Σβόμποντα. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή της, σας. Για τη συνδιάσκεψη μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα, αποτέλεσμα, τα αποτέλεσματά της δεν ήταν αυτό το οποίο είχαμε προσδοκίσει και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερα από ό,τι αναμέναμε πολλοί από εμά, χωρίς τώρα να μπω σε λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά. Αυτό το οποίο εγώ λυπούμε για αυτό ιδίως είναι το θέμα των της διάδοσης των ε, συμβατικών όπλων. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και εκεί θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να έχουν πιο επικοδομητικό ρόλο. Έρχομαι στη διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι πριν από μερικές ε, συναντήσεις μας και ίσως και στην προηγούμενη θητεία είχατε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ιδιαίτερα ενεργή στο διάλογο με τις χώρες της Μέσης Ανατολής για το θέμα αυτό της δημιουργίας μιας ζώνης ελεύθερης από πυρηνικά όπλα. Επομένως το ερώτημά μου είναι, υπήξατε, ήρθατε σε επαφή με τους Ισραηλινούς προηγουμένως και τονίσατε το θέμα αυτό θα είναι στην ημερησία διάταξη. Γιατί γνωρίζουμε ήδη ότι υπάρχει μια πολύ στεναρή στάση από την πλευρά της Αιγύπτου για το θέμα αυτό και νομίζω δικαιολογημένα και ποια ήταν η αντίδραση του Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι θα τους εξέπλητε κάτι τέτοιο ίσως θα θεωρούσαν ότι οι Αμερικανοί κάποιος άλλος θα εμπόδιζαν να τεθεί αυτό το θέμα στην μεση διάταξη. Αλλά πώς βλέπετε να προχωρούν τα θέματα. Μπορείτε να συνεχίσετε το διάλογο αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο το θεωρεί σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση στους επερχόμενους μήνες ότι δεν θέλουμε να υπάρχει ε, γενικά διασπορά ποινικών όπλων. Θέλουμε να το εξασφαλίσουμε αυτό ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ για το σεμινάριο για τη Μέση Ανατολή. Αν λάβετε υπόψη όλες τις δυσκολίες που έχουμε στη Μέση Ανατολή, όλες τις χώρες στην περιοχή και όλες τις δυσκολίες που έχουμε. Και αν αποθαρρυνθούμε από αυτές τις δυσκολίες, δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να εργαστώ, δεν θα μπορούσα να εργαστώ για τον αφοπλισμό αν δεν ήμουν εκφύσεως αισιόδοξη και πολύ πείσμων. Ωραία. Μπορούμε να πούμε στην εαυτό μας δύσκολο είναι, αλλά θα προσπαθήσουμε. Όταν οργανώσαμε το πρώτο σεμινάριο και ήμασταν οι πρώτοι και οι μόνοι που οργανώσαμε τη συνεδρίαση για τα όπλα μαζικής καταστροφής στα στη Μέση Ανατολή, τον Ιούνιο του 1998, όλοι μου είπαν ότι ήμουν παντελώς τρελή και ότι δεν πρόκειται, δεν πρόκειται να τα καταφέρω. Και όμω, τα καταφέραμε. Έγινε το σεμινάριο και όλες οι χώρες συμμετείχαν, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Όλοι ήταν παρόντες. Δεν είχαμε κανένα διπλωματικό ατύχημα. Αντίθετα, όλοι συμπεριφέρθηκαν πολιτισμένα και οι συζητήσεις ήταν ε, κερδοφόρε, επικοδομητικέ. Όχι μόνο επικοδομητικέ, αλλά και συμμετέχοντε είπαν ότι χρειαζόμαστε περισσότερε συζητήσει και είναι ο μόνο τρόπο για να προχωρήσουμε. Και σα παρακαλούμε, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίστε να παίζετε αυτό το διευκολυντικό ρόλο. Σας καλούμε να το πράξετε. Και μάλιστα εξέφρασαν τη θλίψη για το γεγονός ότι κάποιες άτυπες συζητήσεις μεταξύ αραβικών χωρών και Ισραήλ για τον έλεγχο των όπλων ε, σταμάτησαν και ποτέ δεν ξανάρχισαν. Οι χώρε λοιπόν στην περιοχή βρίσκονται σε ένα διέξοδο. Κάποιο πρέπει να δράσει και να παίξει αυτό το ρόλο του διευκολυντή. Αυτό είναι ο φυσικό μα ρόλο. Γιατί στη δήλωση Βαρκελόνη μα ήδη μαζί με όλου του ε, μεσογειακού εταίρου συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ για μια ζώνη ε, ελεύθερη από όπλα μαζικής καταστροφής. Τώρα έχουμε την ε, διάσκεψη αναθεώρηση ε, για τη μη διάδοση των πυρηνικών. Η δήλωση της Βαρκελόνης είναι η βάση για να συνεχίσουμε το διάλογο με το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ έχει προσυπογράψει αυτή τη δήλωση της Βαρκελόνης. Ακόμη και αν δεν θεωρεί ότι οι αποφάσει για τη μη διάδοση των πυρηνικών είναι δεσμευτικές κανονικά είναι. Αλλά κανείς δεν μπορεί να δεσμευτεί από αποφάσεις οργανώσεων στις οποίες δεν ανήκει, αλλά έχει δεχτεί τους στόχους ε, στην δήλωση της Βαρκελόνης για μια ζώνη ελεύθερη από τέτοια όπλα ε, και επομένως μπορούμε να παίξουμε αυτό το ρόλο. Εν συνεχεία, τι άλλο να σας πω. Δεν είναι επίσημη διάσκεψη, είναι ένα σεμινάριο. Και όταν οργανώσαμε το πρώτο σεμινάριο και όταν άρχισα να μιλάω ε, στην αποστολή του Ισραήλ στις Βρυξέλλες για την διοργάνωση ενός νέου δεύτερου σεμιναρίου, μας είπαν ότι δεν μπορούν να μιλήσουν για όπλα μαζικής καταστροφής και μια, για μια τέτοια ζώνη χωρίς τέτοια όπλα, χωρίς να μιλάνε, χωρίς να γίνεται λόγος και να συνδέεται το θέμα με την ε, περιφερειακή ασφάλεια. Δεν λέω λοιπόν ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. Ε, ξέρω ότι τώρα θα έχουμε περισσότερες δυσκολία σαν την πρώτη φορά. Γιατί τώρα έχουμε αυτές τις εντάσεις, αυτές τις αρέσκειες για την ε, συγκεκριμένη αναφορά για το Ισραήλ ε, στο κείμενο της, ε, της συνθήκης αυτής για την ιδιάδοση, αλλά νομίζω ότι είναι ο καθήκον μας να το κάνουμε. Και ο ρόλος μας, όχι μόνο το καθήκον μας, και ο ρόλος μας. Φυσικά όταν πήγαμε στη Νέα Υόρκη, όλοι ήξεραν, και οι Αμερικάνοι, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες ήξεραν ότι θα ήταν προτιμότερο να μην αναφερθεί το Ισραήλ. Όλοι μας φυσικά είχαμε επαφές με διπλωμάτες του Ισραήλ και ξέραμε ότι αυτή η συγκεκριμένη αναφορά στο Ισραήλ δεν ήταν ευπρόσδεκτη. Καλύτερα θα ήταν να την είχαμε αποφύγει για να είμαστε σε καλύτερη θέση για την εφαρμογή της απόφασης. Αλλά όταν είσαι σε μια διάσκεψη με 189 μέρη, πρέπει να λάβεις υπόψη και τις α, απόψεις των υπολείπων συμμετέχων, συμμετεχόντων, των υπολείπων μερών. Η αναφορά στο Ισραήλ σε αυτό το κείμενο δεν γίνεται με αρνητικό τρόπο, όπως σας είπα. Αντίθετα, είναι θετική. Μιλάμε για τη σημασία της προσχώρησης του Ισραήλ στην συνθήκη αυτή μη διάδοσης. Και η αξιολόγηση τελικά ήταν ότι ο βασικός μας στόχος είναι να περισσώσουμε την ε, συνθήκη μη διάδοσης και να εξασφαλίσουμε μέσω αυτής της ε, διάσκεψης ε, στην υιοθέτηση με συνένεση ενός τελικού εγγράφου αντί να έχουμε την αποτυχία που είχαμε πέντε χρόνια πριν. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν δύσκολες αποφάσεις. Τώρα για τις εντάσεις μεταξύ των χωρών που έχουν πυρηνικά και αυτών που δεν έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μονίμως αυτή η ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως. Έχουμε χώρες που έχουν διαφορετικό καθεστώς. Και επομένω τα συμφέροντά τους δεν συμπίπτουν με τρόπο έτσι, φυσικό και προβλέψιμο με αυτά των χωρών που έχουν άλλες, άλλη κατάσταση. Βεβαίως, πριν τη Νέα Υόρκη καταφέραμε να φτάσουμε σε μια κοινή θέση στο Συμβούλιο Και ίσως υπήρξαν μία ή δύο περιπτώσεις όπου στο πρώτο τμήμα της, συνθήκη, της διάσκεψης ε, εκδηλώθηκαν κάποιες εντάσεις. Αλλά στο αποφασιστικό τμήμα της διάσκεψης, που ήταν το τέλος, νομίζω ότι η συνοχή των κρατών μελών πριτάνευσε και ξεπέρασε τις εντάσεις. μπορέσαμε να παίξουμε ένα ρόλο στην διαπραγματευτική ομάδα ακριβώς γιατί η συνοχή υπήρχε και τα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν πυρηνικά και που συμμετείχαν στην διαπραγματευτική ομάδα έπαιξαν ένα ρόλο πολύ επικοδομητικό. Μπόρεσαν να προτείνουν συμβαστικές λύσεις. Δεν δημιουργήσαν προσκόμματα, αντίθετα. Νομίζω ότι σε αυτή τη ε, διάσκεψη για την αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει μεγενθυμένη. Ο πρόεδρος της ομάδας μας ζήτησε πολύ σωστά προς εμάς για να εκπονήσουμε ένα κείμενο συμβαστικό. Μας αναγνωρίζουν ως γεφυροποιούς. Αυτός είναι ο ρόλος που αποδίδει που ε, αποδίδουν οι υπόλοιποι σε μας. Στην BSI δεν συμμετέχουμε πλήρως. Με τα θέματα που είχαμε στα πλαίσια της διάσκεψης για την αναθεώρηση της συνθήκης, μη διάδοση των πυρηνικών, είχαμε πάρα πολλά να κάνουμε. Έχουμε την Σύνοδο Κορυφής ε, για την Πυρηνική Ασφάλεια. Δεν είχαμε χρόνο για, το... για την πρωτοβουλία ειρηνή και ασφάλειας. Τώρα, για την δυσαρέσκεια που εξέφρασε. Ξέρετε ότι κανένα δεν ικανοποιείται ποτέ σε αυτά τα θέματα 100%. Ούτε εγώ. Και όλοι ενδιαφέρονται για τον πυρηνικό αφοπλισμό επίσης δεν είναι 100% ικανοποιημένοι. Όσοι θέλουν ένα καθεστώ πιο έντονο για τη μη διάδοση και αυτοί δεν είναι ικανοποιημένοι 100%. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τα ρίξετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, το θέμα των τακτικών πυρηνικών όπλων. Αναφερόταν στην κοινή μας θέση. Και σας λέω, αν δεν είμαστε πιο φιλόδοξοι και αν δεν πετύχουμε στο σχέδιο δράσης κάτι καλύτερο για τον αφοπλισμό, μάλλον δεν το καταφέραμε αυτό, όχι γιατί δεν είχαμε εμείς ε, ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γιατί τα άλλα κράτη που έχουν πυρηνικά μη, και που δεν ανοίξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλαν καθόλου να γίνει λόγος για τα τακτικά πυρηνικά όπλα. Παρότι εμείς είχαμε λοιπόν ένα κείμενο για τα τακτικά πυρηνικά όπλα, δεν έκανε διαφορά τελικά. Γιατί υπάρχει ε, στεναρή αντίδραση από άλλες χώρες. Δεν μιλάω για τι ευρωπαϊκές χώρες και δεν μιλάω καν για την Αμερική, γιατί τι είπα. Για τις διαβεβαιώσεις ασφάλειας. Δεν συμφωνώ μαζί σας, γιατί τα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν πυρηνικά έχουν δώσει τέτοιε διαβεβαιώσει και έχουν αναγνωρίσει, και αυτό έχει αναγνωριστεί σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία. Και δεν πρέπει να βασιστούμε σε αυτό που κάνει η Κίνα. Αυτό που κάνει η Κίνα είναι ότι δήλωσε ε, ότι δεν πρέπει να κάνει πρώτη χρήση. Που είναι περί περιττό. Γιατί αν έχετε πυρηνικά όπλα, και εγώ δεν προέρχομαι από χώρα που έχει πυρηνικά, αλλά αν έχετε πυρηνικά όπλα, ο μόνο σκοπό του είναι η αποτροπή. Αν δηλώνει λοιπόν ότι πρώτος ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ε, τα όπλα αυτά, τότε καλύτερα ο αφοπλισμό. Αλλά η Κίνα είναι υποκριτική. υποκρίτη παντελώ. Και, λέει, εμεί δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε πρώτα τα πυρηνικά. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να παράγει χάσιμο υλικό. Και είναι αντίθετη στο, στην απαγόρευση χάσιμου υλικού για στρατιωτικού λόγου. Επομένω, αυτό που μου πιο πολύ εμένα είναι το θέμα του σχάσιμου υλικού. Το επιπρόσθετο πρωτόκολλο, προπόθεση για την μεταφορά. Το προτιμούμε. Αλλά στην διάσκεψη αναθεώρηση ήμασταν 189 χώρε, όπω σα είπα. Το καλύτερο που μπορούσαμε να πετύχουμε ήταν το κείμενο που σα διάβασα. Υπάρχει τουλάχιστον κάποια κίνητρα για να το εφαρμόσουμε εν αναμονή της εφαρμογής εν αναμονή τη θέση σε ισχύ μάλλον. Το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό που πετύχαμε επίσης για τις αναφορές. Δεν θέλουμε αναφορές κάθε 6 μήνες. Ο αφοπλισμός και η διάλυση των πυρηνικών ε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ περιπλοκό και τεχνικά και οικονομικά. Το να έχουμε αναφορέ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα δεν έχει νόημα νομίζω. Επίσης, υπάρχει μια πρόσκληση προς τα κράτη που έχουν πυρηνικά για να συμφωνήσουν για ένα συγκεκριμένο έντυπο στις αναφορές σε συγκεκριμένα, με μια συγκεκριμένη συχνότητα, ανατακτά διαστήματα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πρόοδος στο θέμα του reporting των αναφορών. Νομίζω το, το σχέδιο δράσης στον τομέα, στο τμήμα του που μιλάει για τον αφοπλισμό είναι πολύ καλό. Είναι το, το ισχυρότερο σημείο του κειμένου. Αλλά είναι μια διαδικασία, έτσι. Έχουμε μπει σε μια τροχιά και είναι ε, ίσως όπως και ο εμπλουτισμός. Άπαξ και αρχής ο εμπλουτισμός επιταχύνεται. Τώρα, Θέλουμε να υπευθυνοποιήσουμε και τις χώρες όχι μόνο που έχουν ε, επικυρώσει τη συνθήκη, αλλά και τις υπόλοιπες. Υπήρχαν χώρες οι οποίες ήταν κατά, μεταξύ των οποίων και η Κίνα. Για τη συνθήκη απαγόρευση των δοκιμών. Θέλουμε συνένεση λοιπόν για αυτό το θέμα. Αν υπάρχει συνένεση θα σημειωθεί πρόοδος. Το συνολικό αποτέλεσμα όμως είναι πολύ καλό. Σήμερα το πρωί είχαμε την Επιτροπή α, Πολιτικής και Ασφάλειας με τους διαπραγματευτές Ρωσίας και ΙΠΑ που είπαν ότι θεωρούν ότι η έκβαση για τη συνθήκη απαγόρευσης των δοκιμών είναι πολύ θετική. Τώρα έχουμε μια ένα θετικό συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι δυτικές χώρες και οι χώρες που έχουν πυρηνικά μπορούν να συμφωνήσουν πάνω σε ένα κείμενο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε. Είναι το καλύτερο επίτευγμα της Νέας Υόρκης υπάρχει, δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα σύγκληση μεταξύ των διαφόρων υπήρων, μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών ομάδων, μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ευχαριστούμε πολύ για τις δύο αυτές παρουσιάσεις ε, της πλήρης. Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως ε, και πάλι να αναφερθούμε στα θέματα αυτά, ειδικότερα στο θέμα του Ιράν, κατά τους επερχόμενους μήνες. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας, αλλά σε δύο λεπτά. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα δύο λεπτών. Euh, λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα. Περνάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Ενέργειας, Έρευνας και Βιομηχανίας σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης Μέσω Δορυφόρου, αντιμετώπιση των προκλήσεων μελλοντικές δυνατότητες χρηματοδότησης. Τα θέματα αυτά τα έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, αλλά η κυρία Κοπά, η συγγήτρια τη γνωμοδότηση, δεν είχε την ευκαιρία να εκφραστεί στο παρελθόν. Τη δίνω λοιπόν το λόγο τώρα και να μα πει την άποψή τη για τι 10 τροπολογίε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης, συγκεκριμένα το πρόγραμμα Έγνωση και Γαλιλαίο. Η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθυστέρησε και αναμένεται να ανακοινωθεί στις 28 Ιουλίου. Η κατεξοχήν αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΙΤΡΕ, άλλαξε το χρονοδιάγραμμά της για την υιοθέτηση της έκθεσης. Δικός μας ρόλος εδώ είναι να εξετάσουμε τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τις επιπτώσεις του συστήματος Γαλιλαίου για τις διεθνείς σχέσεις και καθώς δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό, ακολούθησα την εισήγηση της Γραμματείας να προχωρήσουμε εμείς κανονικά με την υιοθέτηση ε, αυτής της γνωμοδότησης σύμφωνα με το δικό μας χρονοδιάγραμμα στην Επιτροπή. Πρόθεση της γνωμοδότησης είναι να υπογραμμίσει τη σημασία του Γκαλιλαίου για την ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη συνεργασίας με όλες τις άλλες δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης, ώστε να εξασφαλίσουμε συνέργειες στον τομέα της τεχνολογίας του διαστήματος, αλλά και συμβατότητα και αν είναι δυνατόν και διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Όπως γνωρίζετε, μετά την υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας, η διαστημική πολιτική αναβαθμίζεται και μαζί αναβαθμίζεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συμμετοχή του στην νομοθετική διαδικασία είναι σημαντικό λοιπόν σε αυτή τη γνωμοδότηση να επιβεβαιώσουμε ότι το Galileo is a civil system under civil control χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι ορισμένες τουλάχιστον υπηρεσίες του όπως για παράδειγμα οι λεγόμενες public regulated services είναι διπλής χρήσης και η επιτροπή πρόκειται να υποβάλει την πρότασή της σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης σε αυτές εντός του μηνός. η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας είναι που καταδεικνύει την ανάγκη να μπουν άμεσα κάποια κριτήρια. για παράδειγμα πρέπει να είναι σαφές ότι όλοι οι χρήστες του συστήματος πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο τον καταστατικό χάρτη και τις επιμέρους συμβάσεις του οηε καθώς και τις αρχές που διέπουν τις συνθήκες ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την εξωτερική δράση. δεδομένου επίσης ότι υπάρχουν ήδη τεχνικές δυνατότητες για να αποκλειστεί η χρήση του συστήματος για παράδειγμα για την καθοδήγηση και εκτόξευση πυράβλων ζητάμε από την ευρωπαϊκή επιτροπή ως υπεύθυνη αρχή διαχείρισης να καθορίσει τα απαραίτητα αυτά τεχνικά κριτήρια σε σχέση με τους υποκατασκευή δορυφόρους αλλά και ανησυχίες μας στη διαμόρφωση των κανόνων που πρέπει να διαμορφωθούν σε σχέση με την πρόσβαση στο prs που είναι αποκλειστικής χρήσης των κρατών μελών τα κράτη μέλη θα πρέπει από μέρους τους να συμβάλλουν στην προσπάθεια αναγνωρίζοντας την ευαισθησία του προγράμματος και σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές τεχνολογίες με ιδιαίτερη προσοχή για τα υλικά που αναφέρονται στη σχετική λίστα του διακανονισμού του Βάσεναρ. Τέλος, καθώς το νομικό πλαίσιο είναι ακόμα ισχνό, επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στις προσπάθειες για περαιτέρω εξέλιξη και κωδικοποίηση του διεθνούς δικαίου του διαστήματος. Αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που να δυναμώνει την ήδη αναγνωρισμένη υποχρέωση σχετικά με τη μη στρατικοποίηση του διαστήματος, αλλά και να λαμβάνει δεόντως υπόψη την ευθύνη μας σε σχέση με τα θράψματα και τους εγκατελειμμένους δορυφόρους. Η περιβαλλοντική αυτή διάσταση πιστεύω ότι είναι σημαντική και πιστεύω ότι πρέπει να την αναδείξουμε. Να πω δύο λόγια για τις τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί. Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Ε, τις έχω λάβει υπόψη μου σοβαρά, αν και ορισμένε δεν να, μπορώ να τις αποδεχτώ, γιατί κατά την άποψή μου είναι αντίθετες με το πνεύμα του κειμένου. Τροπολογίες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές είναι η τροπολογία 2, εκδοχή που λέει να ζητάμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε φορά που γίνεται χρήση. Αυτό είναι μη ρεαλιστικό και στερεί τη δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αριθμός 4 είναι σημαντικό για μας να μην χάσει η Ένωση τη δυνατότητα χρήση του Γαλιλαίου, πράγμα που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση Φων Βογκάου η τροπολογία 6. Το ζήτημα της χρηματοδότησης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αναφορά σε supremacy of control in space είναι κατά την εκτίμησή μου υπερβολική. Η 7 που αναφέρεται στην αντίθεσή της για χρήση του Γκαλιλαίου από τις ευρωπαϊκές αποστολές και η 9 που είναι ακριβώς αντίθετη από τη δική μας θέση και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η τροπολογία ένα του κύριου Μπουτίκοφερ μπορεί να γίνει δεκτή, αν και νομίζω ότι το ζήτημα δεν άπτεται άμεσα ζητήματα ασφαλείας και θα το έβλεπα περισσότερο στη σφαίρα αρμοδιότητας της ήτρε ή της ε, επιτροπής προϋπολογισμού. παρ' όλα αυτά δεν δημιουργεί κανένα μείζον πρόβλημα για να περιληφθεί στην έκθεση. όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες νομίζω ότι συμβάλλουν θετικά στην ενίσχυση του περιεχομένου της γνωμοδότησης αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοπά. Ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τη σκιώδη εισηγητρία μας εδώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κοπά για τη γνωμοδότησή της και είμαι σχεδόν απόλυτα σύμφωνος με τις συστάσεις σας σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες. Για την τροπολογία 1 εγώ συμφωνώ επί της ουσίας για αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μπουτικόφερ, αλλά ίσως αυτή η τροπολογία θα πρέπει να πάει στην κύρια έκθεση και όχι στην γνωμοδότησή μας. Αν οδηγήσει στην απόρριψη της γνωμοδότησής μας, τότε θα πάει χαμένη αυτή η τροπολογία. Ίσως σε κάποια άλλη στη θέση να την ε, θέσει ή κάποιο άλλος συνάδελφος στην κύρια επιτροπή να την καταθέσει αυτή την τροπολογία θα ήταν υποφελέστερο. Επίσης, συμφωνώ να απορρίψουμε την τροπολογία 2 και απορρίπτουμε και εμείς όλες τις τροπολογίες της ΓΚΟΕ, δεν συμφωνούμε στην ουσία τους αλλά υποστηρίζουμε την τρία της κυρίας Γκόμης. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι έχω καλύψει τις τροπολογίες από την πλευρά του ΕΛΚ. Αυτή είναι η θέση του ΕΛΚ λοιπόν μπορώ να σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριος Κόφερ. αυτό. Είναι φυσιολογικό που λέτε κύριε Γκάλερ να υποστηρίζετε τις τροπολογίες σας. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό εξάλλου. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 1 τώρα. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από αυτά που είπατε να κάνουμε το, αυτό το οποίο είπατε, να την περιλάβουμε στην κύρια έκθεση να υπάρξει λοιπόν μια τροπολογία, μια υποστήριξη από όλε τι πολιτικές ομάδες για να περιληφθεί στην κύρια έκθεση, εφόσον δεν έχουμε καμία αντίρρηση επί τη ουσία. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 2, θα ήθελα να σας παραπέμψω σε ένα έγγραφο της γερμανικής Bundestag που πρόκειται από μια προφορική ερώτηση το Μάιο του 2010, είναι η ερώτηση 9. Σε ποιο βαθμό βλέπει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τις καθαρά πολιτικές χρήσεις του συστήματος αυτού ότι θα πρέπει να βασίζονται σε κωδικοποίηση του, συστήματος, του, του, συνιάλου του, που αποκλεί την στρατιωτική χρήση και κατά πόσο η PRS, η Public Regulated Service, εξακολουθεί να είναι συμβατή με άλλους χρήστες δορυφορικών σημάτων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα το πρόβλημα της στρατιωτικής χρήσης του συστήματος αυτού. Εδώ είναι το σημείο από το οποίο ξεκινώ από την τροπολογία 2. Δεν λέει η τροπολογία 2 ότι κάτω από όλες τις συνθήκες <clears throat> θα πρέπει να αποκλειστεί η χρήση του συστήματος PRS και στα πλαίσια στε επιχειρήσεων για την διατήρηση της ειρήνης στα πλαίσια ενεργειών της ΚΕΠΑ Απλώς λέει ότι θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να υπάρχει έλεγχος κοινοβουλευτικός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρχει η διευκρίνηση των περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα. Νομίζω και οι δύο στάσεις τίνουν προς τα άκρα. Η μία λέει να χρησιμοποιείται χωρίς κανένα περιορισμό και για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Η άλλη άποψη λέει σε κάποια περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς στόχους αυτό το σύστημα και το περιεχόμενο της τροπολογίας 2 είχε σαν στόχο να υπάρξει κάποιος κανόνας ο οποίος θα οδηγήσει και σε κάποιο μεσαίο δρόμο και ο οποίος να εμπλέκει και να λαμβάνει σοβαρά την ευθύνη και του Κοινοβουλίου για τον έλεγχο του συστήματος αυτού. Γι' αυτό εγώ θα, θα χαιρόμουν αν μπορούσε να μας πει η κυρία εισηγήτρια αν θα μπορούσε να προκύψει κάποια συμφωνία μεταξύ μας ίσως με κάποια διαφορετική διατύπωση εφόσον το επιθυμεί. Αλλά για τους λόγους που ανέφερα και για τους λόγους ε, αυτής της απάντησης που δόθηκε στην Bundestag θα μου ήταν πολύ σημαντικό να βρεθεί κάποια λύση. Έχω ακόμα ένα ερώτημα για την διαμάχη σε σχέση με τις ραδιοσυχνότητες με την Κίνα. Δεν ξέρω κάποιος αν μπορεί να δώσει μια απάντηση για το ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα σε σχέση με αυτή τη διαμάχη για τη χρήση των συχνοτήτων του ραδιοφάσματος. Ευχαριστώ. πολύ. Προτείνω να ολοκληρώσουμε την ε, συζήτηση για τις τροπολογίες και να δώσουμε και το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αν ε, υπάρχει κάτι νεότερο. Η κυρία Λόζινγκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κοπάτνη την Νομίζω ότι έχετε κάνει μεγάλες προσπάθειες για να υπάρξει μια ισορροπημένη γνωμοδότηση στο θέμα αυτό. Και έχετε τονίσει ότι πρέπει να έχει πολιτικό χαρακτήρα το σχέδιο Γαλιλαίο και να μην οδηγήσει σε στρατιοκοποίηση του διαστήματος. Εγώ το υποστηρίζω αυτό απόλυτα, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μου φαίνονται αντιφατικά και κατά την άποψή μας και λαθασμένα ενδεχομένω. Οι προτάσεις σας συγκεκριμένα σε σχέση με τη χρήση του Γαλιλαίου για ε, δράσεις ε, ΚΕΠΑ και για την προστασία κέριων υποδομών. Αυτό είναι για μας μία αντίφαση με τον πολιτικό χαρακτήρα που εσείς έχετε τονίσει στην αρχή της παρέμβασής σας. Εάν χρησιμοποιηθεί ο Γαλιλαίος για την προστασία κέριων υποδομών, κατά τη δική μου εκτίμηση, αυτό δεν σημαίνει αποστρατικοποίηση, αλλά στρατικοποίηση, κάτι το οποίο εσείς έχετε απορρίψει. Στρατικοποίηση στο διάστημα που θα ενισχυθεί με την προστασία αυτών των υποδομών. Είναι απόλυτα κατά η Γκουε μιας στρατιωτικής χρήσης του Γαλιλαίου κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες υπάρχουν ήδη πολύ σημαντικές ε, επενδύσεις στο σχέδιο αυτό, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα σχέδια για στρατιωτικούς λόγους. Εμείς πιστεύουμε ότι στην περίπτωση του Γαλιλαίου θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα πώς θα αποσύρουμε κάποια μέσα από το Γαλιλαίο αντί να προσθέσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για πιο χρήσιμα θέματα όπως είναι παραδείγματος χάρη για κοινωνικές ενέργειες και θέματα ανάπτυξης. Φοβόμαστε λοιπόν ότι ο ελαίος θα οδηγήσει σε κούρσα εξοπλισμών στο διάστημα και στατικοποίηση και γι' αυτό έχουμε καταθέσει τις τροπολογίες μας και θεωρώ ότι μέσω των τροπολογιών αυτών είναι σαφές ότι εμείς κάποιες από αυτές θα τις υποστηρίξουμε ενώ κάποιες άλλες των άλλων κομμάτων δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Merci, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέλλερ. Ίσως δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση συντηρητικοί Γερμανοί βουλευτές εδώ όπως και στην Bundestag. Δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτό που ανέφερε ο κύριος Μπουτικόφερ. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με τη συνθήκη. Η Κομισιόν μπορεί βάσει της συνθήκης να απορρίψει να υπάρξει κοινοβουλευτικός έλεγχος σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα για το πώς θα παρουσιάσουμε αυτό το αίτημα. Νομίζω ότι είναι σαφή η συνθήκη για το σημείο αυτό του ενδεχόμενου κοινοβουλευτικού έλεγχου. Τώρα, για το αν η προστασία των ε, κριτικών των κρισίμων υποδομών αν αποτελεί μια στρατικοποίηση, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν τίθεται έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καθορίζουν τα κράτη-μέλη ποιε είναι οι κρίσιμε υποδομέ και επομένω δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια στρατικοποίηση σε αυτή την περίπτωση. Για μας είναι σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε την τροπολογία αυτή την δύο, θέλουμε να την απορρίψουμε. Merci, Monsieur Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πιστέψτε με ότι δεν είναι από ελληνική αλληλεγγύη ε, που θα συγχαρώ την ε, κυρία Κοπά για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει σε αυτή τη γνωμοδότηση. Άλλωστε τα πολιτικά μας κόμματα βρίσκονται σε οξία πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορώ παρά να εκτιμήσω την ποιότητα της εργασίας που έχει γίνει ε, και να πω ότι συμφωνώ με, την, με όλο το πνεύμα που έχει αυτή η γνωμοδότηση. Ε, θα ήθελα μόνο και γι' αυτό κυρίως ζήτησα το λόγο να αναφερθώ στο κατά πόσο θα γίνεται πολιτική ή κατά κάποιο τρόπο, όπως ακούστηκε, στρατιωτική χρήση ε, του Γαλιλαίου και, εν πάση περιπτώσει, ε, ότι μπορεί να είναι ένα πρόκλημα στρατικοποίησης του διαστήματος. Είναι βέβαιο, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, ότι η ΚΕΠΑ κάνει και civil και military crisis management. Μεγάλο μέρος της ΚΕΠΑ αφορά, μάλιστα, την πολιτική διαχείριση κρίσεων. Επομένως, το να μπορεί τον Γαλιλαίο να αξιοποιείται από τη CFSP με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει στρατικοποίηση ή χρήση του για αμυγό στρατηγικούς σκοπούς. Αισθάνθηκα ότι έπρεπε ε, να, να, τουλάχιστον να παρουσιάσω αυτή την άποψη για να μην υπάρχουν παρανοήσεις ως προς τη χρήση ε, του συστήματος. Και κατά τα άλλα νομίζω ότι η συζήτηση για την συγκεκριμένη γνωμοδότηση θα είναι πολύ σύντομη, διότι δεν έχει και πολλά, να πει κανείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, συμφωνώ απολύτως ε, με όλα αυτά που μόλις είπατε. Μερικές φορές ε, μου κάνει εντύπωση ο υπερβολικός χαρακτήρας ε, αυτής της ε, απειλής της στρατιωτικοποίησης, μιλάμε για ΚΕΠΑ ε, και η μεγάλη πλειοψηφία, δεν νομίζω να αλλάξει αυτό, των ε, αποστολών διαχείρισης κρίσεων είναι πολιτικού χαρακτήρα και ίσως θα πρέπει να δούμε ότι από στρατηγικής απόψεως ε, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, είναι αμερικανικά, τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να μας τα κόψουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή το GPS μπορεί να μην υφίσταται αν θεωρούν οι Αμερικανοί ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Άρα δεν αφορά μόνο στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και, τους, ε, ε, και τις αστυνομικές δυνάμεις ε, που δεν θα μπορούν καν να χρησιμοποιήσουν δορυφορικά, δορυφορικές υπηρεσίες. Κυρία Κοπά, θέλετε να πάρετε το λόγο. Α, πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα μα δώσει πληροφορίε. σε σχέση με την Κίνα. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφός μου καλύτερα, ο Ζερεμί Γκοντέ να τα πει γιατί έχει πρωτοστατήσει στις συζητήσεις με τους Κινέζους και καλύτερα να, μας, να, σας, τα να σας τα πούνε οι πιο αρμόδιοι. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τους Κινέζους, κάναμε πρόοδο τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και γραπτός ε, υπήρξε η αναγνώριση ε, της ε, υπεροχής των συχνοτήτων του ραδιοφάσματος του από σε σχέση με το κόμπας και με όλες βέβαια τις συνέπειες που σημαίνει αυτό για τις ευρωπαϊκές επικοινωνίες. Θα συναντηθούμε μία ακόμη φορά στις 8 και 9 Ιουλίου, τότε είναι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων και είναι σαφές ε, ότι ε, οι Κινέζοι θέλουν ε, αυτή την ρυθμιστική προτεραιότητα να την ανατρέψουν γιατί προτιμούν το δικό του σύστημα από τον Γαλιλαίο. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια κούρσα ανάπτυξης μεταξύ της Ευρώπης και της Κίνας ε, και ε, αυτός που θα αναπτύξει πρώτος το πρόγραμμά του είναι αυτός που έχει την καλύτερη θέση διαπραγμάτευσης, έχει ε, μια προνομιακή θέση διαπραγμάτευσης των ε, ραδιοσυγνωτήτων. Είναι πολύ λοιπόν δύσκολη η κατάσταση, πολλές παράμετροι επισέρχονται και συγκεκριμένα και ε, αφορά και μία από τις παραγράφους της ε, γνωμοδότησης της κυρίας Κοπά, η καλή θέληση των κρατών μελών να μην εξάγουν ευαίσθητες τεχνολογίες που βοηθούν την Κίνα να κατασκευάσει αυτό το, το σύστημα. Αυτό αναφέρεται σε κάποια παράγραφο της γνωμοδότησης του του λεχθέντος. Η άποψή μου είναι ότι σημειώσαμε σημαντικές πρόοδους ε, σε σχέση με την Κίνα, ότι η τάση που αναγνωρίζεται και από τις δύο πλευρές είναι ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία, είναι προς όφελος όλων και προς όφελος των Κινέζων. Ε, ε, για λόγους παρουσίας της Κίνας ε, στο ε, GNSS και για να υπάρξει λοιπόν συμμετοχή της πρέπει να υπάρξει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλους παρόχους συστημάτων όπως το GPS για παράδειγμα και ελπίζουμε να υπάρξει συμφωνία. Έχουμε όμως ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας για τις διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε και νομίζουμε ότι θα είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις ε, για τις οποίες πρέπει να έχουμε μια πολύ συντονισμένη και συνεπή προσέγγιση από πλευράς Ευρωπαϊκή θέσης για να μην χάσουμε έδαφος διαπραγματεύσεις Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι σε σχέση με τη χρήση του Γκαλιλαίου για τις ε, αποστολές ε, ΚΕΠΑ και τη χρήση ε, του GPS του Αμερικανικού. Δυστυχώς δεν έχουν όλες οι χώρες ευρωπαϊκή Ένωση το GPS του Αμερικανικό, δεν έχουν την ίδια πρόσβαση. Υπάρχει και μία εξάρτηση συνεπώ από το GPS. Με τον Γαλιλαίο όμως ε, τα κράτη-μέλη θα έχουν τα ίδια μέσα, την ίδια πρόσβαση και επομένως ε, τα πράγματα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνοχή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Λόζινγκ θέλει να πάρει το λόγο. Μια μικρή διευκρίνηση ακόμα. Ο κύριος Φερχόγγεν στο παρελθόν είχε πει ότι ο Γαλιλαίος είναι πρόγραμμα με μεγάλη στρατιωτική ε, ε, χρησιμότητα. Εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον που πρέπει να σας το υπενθυμίσει ένα μέλος της ΓΚΟΕ αυτό. Ε, Κυρία Κοπά. Πρόεδρε, μία λέξη γιατί βλέπω ότι έχει περάσει πολλές, ε, πολλή ώρα ε, ο γκαλιλαίο μπορεί να εξασφαλίσει την αυτονομία της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανεξαρτησία της. δεν είμαστε εναντίον της στρατικοποίησης αλλά δεν πρέπει να έχουμε μια σχέση ενοχής σε σχέση με τις αποστολές της κοινή ε, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. σκεφτείτε την επιχείρηση αταλάντα και το ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει το γαλιλαίο σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και συνολικά για όλα τα θέματα διαχείρισης κρίσεων. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα μπρος για την ε, ε, Ευρώπη και γι' αυτό ε, αξίζει να το στηρίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ο κύριος Μπουτίκοφερ, για τον κύριο Μπουτίκοφερ άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τα σχόλιά του για την τροπολογία 2. Με μεγάλη ευχαρίστηση θα περιμένω μια διαφορετική διατύπωση ώστε να τη συζητήσουμε μήπως μπορεί ε, να γίνει αποδεκτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα υιοθετήσουμε αυτή τη γνωμοδέτηση. Θα ψηφίσουμε στην ΑΦΕΤ ε, στις 22-23 ε, Ιουνίου. Και τώρα μας πιέζει ο χρόνος. Mm. Περνάμε στο σχέδιο πρότασης για ένα κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογία διπλή χρήση. Ο συντάκτη ε, του σχεδίου γνωμοδότησης είναι ο κ. Μπουτίκοφερ. Έχει το λόγο. Um, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Είναι προβληματικό το ότι πιέζομαστε τόσο πολύ από το χρόνο. Αυτό το θέμα δεν είναι απλώς τεχνικό, είναι εξόχως πολιτικό. Ζητώ λοιπόν την κατανόησή σας για να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω ένα-δύο ανθρώπους που με βοήθησαν για να συντάξω την εκνομοδότηση, ιδίως α, το Μιχάλ Μανολιόβιτς από τη Γραμματεία, τη Ρόσμαρη Χαμπάνσκι από το Συμβούλιο και τον κύριο Γουισκόφσκι από την ε, Κομισιόν. Με βοήθησαν και με διαφώτισαν σε πολλά σημεία. Εγώ αντιμετωπίσω αυτό το, θέμα από τη σκοπιά της ασφάλειας και της ειρήνης. Αυτό είναι το καθήκον μας. Φυσικά, η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η ΙΝΤΑ, Διεθνούς Εμπορίου. Αυτοί έχουν διαφορετική προσέγγιση. Εμείς όμως θα πρέπει να εστιάσουμε σε θέματα ασφάλειας. Γενικώ πώς. Θέλω να σας πω ότι Προτιμώ τη στάση του Συμβουλίου για αυτά τα θέματα και όχι τη στάση της Επιτροπής. Το Συμβούλιο στις συζητήσεις για την πρόταση εστίασε στα μελήματα περί ασφάλειας, πολύ περισσότερο από την Κομισιόν. Η άποψή μου και η γνωμοδότησή μου ε, συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με τις ιδέες που εξέφρασε το Συμβούλιο. Δεν πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει δίκιο όταν μιλάει για αυτά τα είδη της χρήσης και τα χαρακτηρίζει ως μη ευαίσθητα. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα η ε, έτυχε επίθεσης ο οικονομικός ε, σχεδιασμός και ο όρος πόλεμος δεν είναι κατά τύχη ψηλά στην ατζέντα του ΝΑΤΟ για την αναθεώρηση της, ε, των στρατηγικών, της στρατηγικής θεώρησης. Επομένως, τέτοια θέματα θα πρέπει να τα λαμβάνουμε πραγματικά υπόψη. Δεύτερον, η Κομισιόν προσπαθεί να προτείνει κάποιες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής της, χωρίς να είναι σε θέση να μας λέει, μέχρι τούδε τουλάχιστον, πώς πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι προϋποθέσεις. Αντίθετα τώρα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στις ΗΠΑ έχει μερικές χιλιάδες υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους που ελέγχουν την εξαγωγή ευαίσθητων ειδών σε συγκεκριμένους προορισμούς. Ποιος θα τα κάνει αυτά εδώ στην Ευρώπη, ποιος θα το κάνει αυτό το, αυτόν τον έλεγχο, μήπως η τελωνιακή, στα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό εδώ. Με βάση αυτά που προτείνει το Συμβούλιο επίσης, δεν θα πρέπει να δώσουμε άδειε στις εξαγωγές για είδη χαμηλής αξίας. Έχω προτείνει διάφορες τροπολογίες για τη γενική άδεια εξαγωγών η οποία θα ισχύει ούτως ή άλλως αυτή η γενική άδεια. Αλλά από τη σκοπιά της ασφάλειας είναι σωστό να λέμε ότι οι περιορισμοί που τα επιμέρους κράτη-μέλη έχουν επιβάλει στο παρελθόν δεν θα πρέπει να αγνοηθούν. Ας μην εφαρμόσουμε την πιο επίκη, την πιο ελαφριά αν θέλετε αντιμετώπιση, την πιο χαλαρή λύση που έχουν βρει ποτέ τα κράτη-μέλη. Ας λάβουμε ως κοινό παρανομαστή την πιο προσεκτή και την πιο αυστηρή στάση που είχαν τα κράτη-μέλη και αυτή να τη χρησιμοποιήσουμε ως κανόνα. Ούτως ώστε να υπάρχει μια εναρμόνιση. που δεν θα υποσκάψει το επίπεδο ασφάλειας κανενός κράτους μέλους, ούτε του πιο αυστηρού. Αυτή είναι η γενική φιλοσοφία. Και κάτι ακόμα. Τελευταίο. Θέλω να υπάρχει μια συνετή στάση, μια συνετή προσέγγιση. Γιατί δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Δεν έχουμε στοιχεία για την τελική χρήση αυτών των ειδών διπλής ε, χρήσης που εξάγονται από την Ένωση. Στο βαθμό που δεν έχουμε αυτά δεδομένα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πορευτούμε συνετά, όπως είπα. Τώρα, δεν θα διατρέξω τις επιμέρους τροπολογίες που σας προτείνω. Υπάρχει και ένα πρόβλημα τύπων η Ισπανική Προεδρία δεν μας ε, μοίρασε ένα κείμενο της Προεδρίας. Και το κείμενο εργασίας μας είναι ούτως ή άλλως ξεπερασμένο από τα γεγονότα. Είναι παράδοξο που η υποεπιτροπή μας πρέπει να συζητάει βάσει κειμένων που δεν είναι επικαιροποιημένα. Δεν προτείνω να αυτά την αναβολή της ψηφοφορίας για τις τροπολογίες, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση επιζήμια για μας, να μην ληφθεί υπόψη δηλαδή η δική μας γνώμη. Καθόλου. Δεν θέλω κάτι τέτοιο. Θέλω να πούμε όλοι μας ξεκάθαρα όμως και να αναγνωρίσουμε ότι το Κοινοβούλιο εργάζεται μέσα σε δύσκολες συνθήκες και δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα ούτως ή άλλως ε, στη συνεδρίασή μας της 12ης Ιουλίου, προθεσμία για τις τροπολογίες. ...9 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Προτείνω λοιπόν να μην κάνουμε τη συζήτηση αυτή τη στιγμή... ...εκτός αν κάποιος διακατέχεται από φοβερό πόθο να πάρει το λόγο τώρα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Merci pour... Ευχαριστώ πολύ που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιε παρατηρήσει θα ήθελα να κάνω ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπω κατηγορείται για υπερβολική επίοικια και δεν λαμβάνει επαρκώ υπόψη την πτυχή τη ασφάλεια. Ε, σε σχέση λοιπόν με αυτό που είπε ο εισηγητή ε, για το γεγονό ότι είναι λίγο παροχημένη η πρόταση, θα ήθελα να πω στου παρόντε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα κράτη-μέλη να ενισχύσει τον κανονισμό που αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών ε, με έλεγχο τη διαμετακόμισης όπως επίσης και τη ε, διαμεσολάβηση ε, για την πώληση ή την εξαγωγή όπλων. συγγνώμη, ειδών διπλής χρήσης. ο κανονισμός είναι ο 428 κάθετος 2009. Επομένως, εν μέρη έχει δίκιο ο εισηγητής που λέει ότι από τότε έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και ο κανονισμός στον οποίο βασίζεται η ε, έκθεση έχει μάλιστα αλλάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως είχε προτείνει ακόμη περισσότερες ε, τροποποιήσεις για να ενισχύσει την ασφάλεια και ειδικότερα σε σχέση με τα αγαθά που συνδέονται με τον Γαλιλαίο. Και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος ε, για την εξαγωγή ορισμένων πολύ ευαίσθητων ε, ειδών και τεχνολογίας προς άλλες χώρες. Εμείς ε, δεν, αποφασίζουμε αυτόν τον κατάλογο. Τα κυρίαρχα κράτη-μέλη αποφασίζουν τον κατάλογο των ειδών αυτών και στις περισσότερες περιπτώσεις, διαπραγματεύσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκπροσωπείται καν. Όσον αφορά τώρα οι πρακτικές των μεγαλύτερων εξαγωγέων ε, ειδών ε, τέτοιου είδους, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, Αν δείτε λοιπόν τον κατάλογο των ε, ειδών διπλής ε, χρήσης, θα δείτε ότι έχετε περίπου 200 σελίδες ε, τεχνολογίας που την χάνουν ελέγχου για εξαγωγή προς οποιοδήποτε προορισμό. Επειδή κάποια κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων εξάγουν περισσότερα και έχουν μεγαλύτερη εμπειρία για τη χρήση τη στρατιωτική της τεχνολογίας αυτής και μιλάω για τη διπλή χρήση, δηλαδή για είδη που έχουν να κάνουν με ε, αστική χρήση που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτική χρήση. Μιλάμε για χημικά προϊόντα, για παράδειγμα, για μηχανισμούς, για ε, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για πράγματα που τα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα στην καθημερινή μας ζωή. Πριν από πέντε χρόνια ελέγχαμε και τους υπολογιστές αυτούς τους καταλόγους ε, και μιλάω για τους υπολογιστές που χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εφημερίδων ε, Γι' αυτό λοιπόν ε, οι χώρες ε, που ε, κάνουν πολλές εξαγωγές, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένε Πολιτείες, έχουν ζητήσει τον έλεγχο των εξαγωγών προς συγκεκριμένους προορισμούς σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε ποιες είναι οι τεχνολογίες και ποιες, ποιοι είναι οι προορισμοί και ποιες είναι οι συνθήκες για τις οποίες θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον έλεγχο. Δεν λέω να τον καταργήσουμε τον έλεγχο Απλώ, στο παράρτημα 2 του κανονισμού ε, του ισχύοντος, στον κατάλογο των εξαγωγών, Υπάρχουν κάποιες χώρες που ε, ευνοούν τις εξαγωγές προς χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ε, η Αυστραλία κλπ όλες αυτές οι χώρες είναι μέλη καθεστώτος ελέγχου εξαγωγών και επομένω διέπονται από, τις ίδιες, ε, ε, από τους ίδιους όρους ε, με τα κράτη-μέλη. Οπότε να προσέχουμε λίγο τι λέμε και το λέω αυτό με κάθε σεβασμό προ τον Ευρωβουλευτή. Ο στόχος μας δεν είναι να ε, μην υπάρχει ασφάλεια. Στο παρελθόν, ε, στο πρόσφατο παρελθόν, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εναρμόνιση των ελέγχων στα κράτη-μέλη για τα είδη που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. Δείτε τι έγινε με το Ιράν. Τι υπάρχει στις κυρώσεις για το Ιράν. Υπάρχει ένα τμήμα ειδών που δεν αναφέρονται ε, στο καθεστώς αυτό ελέγχου εξαγωγών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ή να τα καταργήσει ή να τα μειώσει γιατί ένα τμήμα της εξάρνησης των εξαγωγών που, που κάνουν τα κράτη-μέλη αφορούν συγκεκριμένα είδη τα οποία δεν αναφέρονται στον κατάλογο. Και γι' αυτό ακριβώ είχαμε προτείνει και τα σχετικά με τον Γαλιλαίο είδη και τα κράτη-μέλη το αρνήθηκαν αυτό. Και σα το λέω αυτό για να το γνωρίζετε ότι σε αυτές τις πάνω από 200 σελίδες τεχνολογίας υπάρχουν προϊόντα που ελέγχονται, κατά, τον οποίο η εξαγωγή ελέγχεται τα τελευταία 30 χρόνια σε σχέση με τον όγκο των εξαγωγών που είναι περίπου 5 με 10% του ε, συνολικού εμπορίου. Οπότε, 0,5% όλων αυτών των ελεγχόμενων προϊόντων ε, την χάνουν άρνησης ε, εξαγωγών και αυτό ήταν μια προσπάθεια που κάναμε για να μειώσουμε τους κινδύνους και να εναρμονίσουμε ε, την άποψη των κρατών μελών για, ζητήμα, για, ειδικά, για είδη που δεν είναι ευαίσθητα. Όταν λοιπόν το είχαμε προτείνει αυτό, τα κράτη-μέλη δεν είχαν κρίνει απαραίτητο να αρνηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγες παρατηρήσεις. Η δική μου θέση εδώ είναι βασικά η θέση η οποία προέκυψε από μακρές διαπραγματεύσεις μέσα στο Συμβούλιο. Δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ελαφρά την καρδία. Τα θέματα ασφάλειας εξακολουθούν να παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και το Συμβούλιο παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο επομένω. Δεν λέω τώρα ότι η Κομισιόν δεν έχει λόγο στα θέματα ασφάλειας, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Λέω όμως ότι το Συμβούλιο έχει, μεγάλη, έχει διαφορετική προτεραιότητα στα θέματα αυτά. Άκουσα την άποψη της εκπροσώπου της Κομισιόν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις πρακτικές των μεγαλύτερων χωρών εξαγωγέων. Εγώ εκπροσωπώ μία από αυτές τις χώρες, αλλά δεν θα τολμούσα να πω ότι επειδή είμαστε μεγάλη χώρα έχουμε δίκιο. Πρέπει να στηριχθούμε στην αρχή της πρόληψης, της προφύλαξης να ακολουθήσουμε αυστηρούς κανόνες, ότι τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να σεβαστούν τους πιο αυστηρούς κανόνες που έχουμε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί οι χώρες οι οποίες είναι μεγάλη εξαγωγής δεν είναι κατά ανάγκη οι χώρες οι οποίες ενδεχομένως θα υποστούν, θα υπόκεινται σε μεγαλύτερες απειλές αν τα αγαθά διτής χρήσης χρησιμοποιούσαν με καταχρηστικό τρόπο. Υπάρχει το παράδειγμα μια μικρή χώρα η οποία βρέθηκε κάτω από επίθεση στον κυβερνόχωρο. Δεν ήταν μεγάλη χώρα, δεν ήταν χώρα που είχε εξαγάγει υλικό πληροφορική, αλλά υπέστη μεγάλη πίεση. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μέλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα πρότυπα ασφαλείας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο εάν ακολουθήσουμε μια αυστηρή προσέγγιση. Ποιος είναι η αρχή που εξασφαλίζει τον έλεγχο των εξαγωγών. Από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη έχουν ενώπιον τους κάποια πρότυπα, μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη του ελέγχου βάσει αυτών των προτύπων. Τότε δεν θα υπάρχει και δυνατότητα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυστηρότερους κανονισμούς ασφάλειας. Αυτό είναι ακριβώς το, το θέμα. Δεν λέω ότι αυτό δεν είναι μια καλή ιδέα. Δεν λέω ότι αυτή η ιδέα δεν πρέπει να προωθηθεί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε γενική έγκριση των εξαγών. Λέω, αλλά εάν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι νιώθουν ικανοποιημένοι και ασφαλείς. Αυτή είναι λοιπόν η θέση, όχι μόνο η δική μου προσωπική θέση, αλλά και η θέση η οποία προέκυψε στις συζητήσεις στους κόλπους του Συμβουλίου. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα παρακαλώ, γιατί έχουμε και άλλα σημεία στην μέση ένταξη. Κύριε Κόβατσεφ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Συμφωνώ με τον κύριο Μπουτικόφερ ότι η γνωμοδότησή μα θα πρέπει να επικεντρωθεί στα, στα θέματα ασφάλεια και να αφήσει ε, τα θέματα τη βιομηχανία στην ίντα. Η εξαγωγή αυτών των προϊόντων και αυτής της τεχνολογίας ε, εμπεριέχουν ε, υψηλό κίνδυνο και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς. Γι' αυτό αυτά θα πρέπει να ελέγχονται. Δεν ξέρω πώ γνωρίζετε τη θέση του Συμβουλίου, γιατί υπάρχει από ό,τι ξέρω μια ομάδα εργασία ε, στο Συμβούλιο που θα ε, αποφασίσει επί τη πρόταση της Κομισιόν, θα γνωμοδοτήσει δηλαδή η ομάδα του Συμβουλίου στι 11 Ιουνίου. Πώ την ξέρετε εσεί, λοιπόν ήδη τη θέση του Συμβουλίου. Συμφωνώ όμω ότι η κυβερνοασφάλεια ε, έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία μας, ε, η άμυνά μας, ε, όλος ο κρατικός μηχανισμός ε, εξαρτάται πάρα πολύ από τον τρόπο μεταφοράς αυτής της ε, ευαίσθητης τεχνολογίας και της χρήσης της. γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κυβέρνο επιθέσεις. Και αυτό πρέπει να αποφευθεί. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ισορροπημένη και εξασφαλίζει επαρκή προστασία και εγγύησεις για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι που ανέφερα. Φυσικά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία αλλά συνολικά υποστηρίζω την πρόταση τη Κομισιόν. Εγώ είμαι, προέρχομαι από μια κομμουνιστική χώρα και συμφωνώ με τι ανησυχίε του κ. Μπουτικόφερ για την ε, εξαγωγή ειδών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την, το στραγγαλισμό της ε, ελευθερίας σκέψης και την ελευθερία λόγου και τη ελευθερίας λόγου όπως γίνεται στην Κίνα ή στη Ρωσία. Ε, ευχαριστώ που ήσασταν ταχύτατη κυρία Λέζινγκ. Θα είμαι σύντομη η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη θέση του κύριου Μπουτικόφερ. Είναι σαφής λοιπόν η θέση που εξέφρασε ο κύριος Μπουτικόφερ και είναι απαραίτητο να υπάρξουν και να υπάρξει υποστήριξη ορισμένε δικέ μα τροπολογίε, οι οποίε διευκρινίζουν ακόμα καλύτερα αυτήν την ε, θέση. Ο κύριο Έλε. Εμεί έχουμε τεχνικέ δυσκολίε με αυτά που αναφέρονται στις τροπολογίες 16, 17 και 18 που ζητούν απόλυτη διαγραφή των παρατημάτων F και D. Αυτό είναι ένα θέμα ουσίας. Εδώ δεν έχουμε ακόμα τη θέση του Συμβουλίου σε σχέση με ένα θετικό κανόνα. Όταν λέμε <clears throat> υπολογιστές και παρελκόμενα όλα αυτά που είναι στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με μια διτή χρήση δεν μπορούμε να αποκλείσουμε όλους τους υπολογιστές απλώς και μόνο επειδή έχουν δίτη δυνητικά χρήση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπορέσει να καταρτήσει η Κομισιόν ένα θετικό κατάλογο, αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο το Κοινοβούλιο, το οποίο δεν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη, να προβεί αυτό στην κατάρτιση ενός καταλόγου. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα με αυτή τη συζήτηση να διαλευκάνουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, οι τροπολογίες... Α, το Συμβούλιο, αλλά ταχύτατα. Θα ξανασυζητήσουμε ούτως ή άλλως αυτό το θέμα τον Ιούλιο. Και ούτως ή άλλως μας μένουν και άλλα σημεία στη μέση διάταξη, πολύ σύντομα. Η Γραμματεία του Συμβουλίου ε, σημειώνει ότι την πρόταση της Επιτροπής ε, με έναν ε, μακρύ κατάλογο από χώρε και είδη που πρέπει να υποφεληθούν από την άδεια εξαγωγής και Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες ασφαλείας των χωρών μελών, ε, τα είδη που θα συμπεριληφθούν στην άδεια εξαγωγή και ο κατάλογος των χωρών που θα υποφεληθούν από τη Γενική Άδεια Εξαγωγή θα πρέπει να αποφασιστούν από τα κράτη-μέλη ε, στην ομάδα εργασίας για τη διτή χρήση αυτών των ειδών και της τεχνολογίας. 9 Ιουνίου λοιπόν οι τροπολογίε και η επόμενη συζήτηση τον Ιούλιο στις 11 εδώ στην Υποεπιτροπή. Τάχιστα θα περάσουμε τώρα στην αντιπροσωπεία τη ΕΝΤΕ που πήγε στο Northwood την περασμένη εβδομάδα τρία άτομα, η κυρία Σούλη που είναι εδώ, ο κύριος Λουάν ο οποίος δεν είναι, απουσιάζει και ο κύριος Κάμπερ Μπόναμον ο οποίος είναι παρόν. Έχετε το λόγο, Κατρίν. Ε, επισκεφτήκατε το αρχηγείο της ε, επιχείρησης Αταρλάντα της ε, Βρετανικής και Ολλανδικής ομάδας ε, μάχης και το Αρχηγείο Θαλάσσιας ε, Επιχείρησης ε, ε, κατά της πειρατείας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. πολύ πυκνή ημέρα. πρώτη φορά είδα τόσα πολλά αρχηγεία στη ζωή μου στον ίδιο χώρο. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα της καταλληλότητας του να συγκεντρώνται τόσα πολλά αστέρια και γαλόνια στον ίδιο τόπο, αλλά πέρα από αυτή την επιφύλαξη όλα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα γιατί και σε επίπεδο ΝΑΤΟ ε, υπήρχε απόλυτη σύμπνοια γιατί ούτως ή άλλως είναι θαλάσσια επιχείρηση. Νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη σύμπνοια και όλα πηγαίνουν κατευχήν. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί η επιχείρηση Αταλάντα, είναι απόλυτα απαραίτητη ε, για αυτή τη ζώνη. Υποστηρίζει το πρόγραμμα για τον παγκόσμιο επισητισμό, παρότι τελευταία κάποια πλοία δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν λόγω επιθέσεων και γιατί επίσης περνούν από αυτή τη ζώνη εμπορικά πλοία. Ε, τώρα, πιο συγκεκριμένα, πέρα από το 2006, πρέπει να βρούμε το budget για να συνεχίσουμε αυτή την επιχείρηση, αλλά και να βρούμε ε, ποιες είναι οι ρίζες αυτού του κακού. Δηλαδή, να σταθεροποιήσουμε την ε, περιοχή. Παρακαλώ μπορείτε να βγείτε ήσυχα από την αίθουσα. Και αν θέλετε να κάνετε πηγαδάκια εκτός αίθουσα. Να δούμε λοιπόν ποιε είναι οι ρίζε του κακού ε, στην περιοχή. Δηλαδή να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα στη Σομαλία. Αυτά για το πρώτο τμήμα. Πάω πάρα πολύ γρήγορα. Ε, για τις ομάδες μάχης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία. Ε, δεν αναπτύχθηκαν ποτέ όμως μέχρι στιγμής. Κρίμα είναι αυτό και το, και, το λένε και οι διοικητές, θα μπορούσαν αυτές οι ομάδες να υποστηρίξουν ε, πολιτικές επιχειρήσεις και αποστολές. Ε, αυτή η σχηματισμή μάχης λοιπόν. Γιατί οι πολιτικές επιχειρήσεις δεν έχουν αυτή την, αυτό το know-how, αυτή την ε, τεχνογνωσία. Πολύ συνοπτική. Μπράβο σας. Και εγώ βρήκα πάρα πολύ χρήσιμη αυτή την επίσκεψη και θέλω να αποτίσω φόρο τιμή σε αυτούς τους ε, στρατιωτικούς οι οποίοι διευθύνουν τι επιχειρήσεις στο Northwood. Δυστυχώς δεν βρήκαμε τον ε, διοικητή, τον ε, υπονάβαρχο, γιατί είχε να πάει στην κηδεία ενός άλλου στρατιωτικού ο οποίος σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν. Είναι σημαντική η θυσία στρατιωτικών στο Αφγανιστάν. Πρέπει να αποτίσουμε φοροτιμή σε όλους τους στρατιωτικούς που υπηρετούν εκεί εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια παρατήρηση ότι υπήρξε ένα κίνδυνο, ένα θέμα επικάλυψης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της, να, της ε, ναυτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΝΑΦΟΡ, που είναι η πρώτη ναυτική δύναμη που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Ένωση πότε, για το θέμα της ε, Σομαλίας. Ρωτήσαμε το ΝΑΤΟ αν θα είχε νόημα να υπάρχει ενιαία ε, δίκηση για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με, την, με τον έλεγχο της περιοχής και μας είπε ναι, πράγματι ο διοικητής του ΝΑΤΟ θα ήταν πολύ καλύτερα να έχουμε μια ενία διεύθυνση. Και είπε ότι υπάρχουν προβλήματα ότι οι Ηνωμένες, η, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε πληροφορίες και εικόνες από δορυφόρο, κάτι το οποίο δεν βοήθησε την ε, επιχείρηση δεν λέω ότι υπάρχουν προστριβέ μεταξύ των δύο, αλλά τη στιγμή που έχουμε 21 από τα 27 κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο ΝΑΤΟ, υπάρχει το θέμα αυτό τη επικάλυψη των προσπαθειών, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί σε τελική ανάλυση είναι μια πολύ σημαντική αποστολή. Είναι ένα από τα κύρια σημεία ελέγχου στον κόσμο σε ό,τι αφορά τι ναυτικέ μεταφορές και όπου απειλείται η ναυτιλία από την πειρατεία. Η πειρατεία ενός πλοίου οδήγησε στην αύξηση των τιμών πετρελαίου σε όλο τον κόσμο κατά 1,4%. Όλες οι, οι συνέπειες λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Επομένως, το να συνεργαστούμε και να αποφύγουμε την επικάλυψη προσπαθειών αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερο να το κάνουμε μέσα από το ΝΑΤΟ που είναι ένα καλύτερα πεπειραμένο σύστημα γιατί υπάρχει μεγάλη επικάλυψη, είναι τα, <clears throat> τα ίδια πλοία. Τη μια μέρα έχουν τη σημαία του ΝΑΤΟ, την άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο όμως λαμβάνεται υπόψη τακτικά. Κύριε Ταν Νοκ, <clears throat> πάρα πολύ σύντομα ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο Ντέβιτ Κάμπελ. Εγώ θα είχα την ίδια εντύπωση μαζί του στο παρελθόν, αλλά έχω μεταστραφεί. Ήμουνα πρόσφατα στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και θα τα πει αυτά μετά ο κύριος Σαρσβόλσκι, αλλά η δική μου εντύπωση ήταν ότι η ΝΑΒΦΟΡ έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του ΝΑΤΟ. Ακόμα και το ΝΑΤΟ θα το συμφωνήσει αυτό, έστω και με δυσκολία, ότι υπάρχει και κάποια συνεργασία με χώρες που, που είναι αδέσμευτες, όπως είναι η Ινδία, παραδείγματος χάρη, οι οποίες αλλιώς δεν θα συνεργαζόντουσαν με κάποια επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Επομένως, αυτή είναι η αξία που φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την αποστολή και είναι το γεγονό ότι μπορεί να είναι πιο αποδεκτή αυτή η αποστολή από άλλε χώρε και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Σας λέω ότι θα κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση της, της υποεπιτροπής μας για την πειρατεία και την αντιμετώπιση της πειρατείας και θα έρθουν και οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι οι οποίοι θα μας τονίσουν αυτό που είπε ο κύριος ε, Τάνοκ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συνεργάζονται με αυτήν την ε, επιχείρηση έχουν ήδη οι διερμηνείς υπερβούν, υπερβούν το χρόνο, έχουν υπερβεί το χρόνο τους. Αν δεν έχετε αντίρρηση, η έκθεση για την ε, ε κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ μπορούμε να συνεχίσουμε μόνο στα αγγλικά, αν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Όσοι θέλουμε να μην ε, ακούσουμε. Εντάξει. Ή στα γαλλικά. Ε, εντάξει, ό,τι θέλετε. Για να απελευθερώσουμε λοιπόν τις διερμηνείς. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και διερμηνείς.